Um, Γεια σας συνάδελφοι. Θα αρχίσει λοιπόν η συνεδρίαση. Πάμε αμέσω στο πρώτο θέμα, έγκριση μερίσιας διάταξης. Ε, παρακαλώ, για το πρώτο σημείο σημειώστε ότι οι συστάσει των συντονιστών τη 5 η Οκτωβρίου θα σα υποβληθούν προ έγκριση αύριο το μεσημέρι στι 3 η ώρα. Επαναλαμβάνω, ε, οι συστάσει των συντονιστών τη 5 η Οκτωβρίου που ήταν η περασμένη μα συνεδρίαση θα σα υποβληθούν αύριο προ έγκριση στι 3 η ώρα πριν τι ψηφοφορίε ακριβώ. Εάν δεν έχετε αντιρρήσει, εγκρίνεται λοιπόν το σχέδιο τη διάταξη. Λοιπόν, σημείο 2. Ε, διερμηνία κροατικά και εγώ ιδελικά δυστυχώ, σήμερα και αύριο δεν θα έχουμε ε, για τις συστάσεις των ε, συντονιστών με βάση το άρθρο 205 γραπτή διαδικασία ενέκριναν μια γνωμοδότηση υποτύπου επιστολή για την Επιτροπή Προπολογισμού για το διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 7 στον προπολογισμό του 2015 για το μέσο ευελιξία και την κινητοποίησή του για να ανταποκριθεί στην προσφυγική κατάσταση. Ε, σύμφωνα με το άρθρο 205, το εγκρίνεται, το εγκρίνει η Επιτροπή. Επίσης, συμφώνησαν οι συντονιστές να συνεδριάσουμε από κοινού με την Επιτροπή Προπολογισμού για θέματα προσφύγων και μεταναστών στις 19 Οκτωβρίου από τις 18.45 μέχρι τις 20.30 στην αίθουσα Γιάν 6Q2. Σημείο 4. Διεθνείς συμφωνίες. Ενημέρωση σύμφωνα με το άρθρο 210 παρένθεση 10 της Συνδίκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να σας ενημερώσω ότι έλαβα πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου που θα ληφθεί ε, απόφαση από τα σχετικά όργανα για τη συμφωνία με τη ε, Καπβερδιανή Δημοκρατία για ε, την έκδοση θεωρήσεων διαβατηρίων μικρής διάρκειας για σύντομες ε, βραχίες μάλλον Ε, ε και ε, για την ψηφοφορία αύριο θα ψηφίσουμε από τις 3 μέχρι τις 5 παρακαλώ να έχετε μαζί σας τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας σας. And we move to the... Πάμε λοιπόν στο σημείο 3 για τη νομική βοήθεια για ε, υπόπτου ή κατηγορουμένου που στερούνται τη ελευθερία του και τη νομική συνδρομή σε διαδικασίες εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Ε, ο εισηγητή μα είναι ο κύριο Δε Γιόγκ. Εδώ παρόν, η πρόταση οδηγία για νομική συνδρομή για υπόπτου ή κατηγορούμενου που στερούνται τη ελευθερία θα μα ενημερώσει μετά το δεύτερο τριμερή διάλογο τη 29 Σεπτεμβρίου ο εισηγητή κύριο Δε Γιόγκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δέκα λεπτά έχω. Λοιπόν, θα είμαι σύντομο και μπορώ να είμαι και σύντομο, διότι ουσιαστικά δεν καταφέραμε τίποτα ακόμα. Υπό την έννοια αυτή δεν έχω και πάρα πολλά να σα πω. Γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε ζητήσει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογή για την οδηγία. Ε, θα πρέπει ε, να γίνει ε, λόγος για νομική συνδρομή και υπόπτωση κατηγορουμένους που στερούνται της ελευθερία τους, λέει. Νομική συνδρομή θα πρέπει να χορηγείται προς όλους και η οδηγία που δίνει πρόσβαση σε δικηγόρους και συνηγόρους και που εγκρίναμε το προβλέπει αυτό. Δηλαδή σημαίνει ότι υπάρχει σχέση ένα προ ένα με την παρούσα οδηγία και με οδηγία που ήδη ισχύει. Το Συμβούλιο δεν το βλέπει καθόλου έτσι. Ε, το Συμβούλιο ε, θέλει να το περιορίσει ακόμα περισσότερο και δεν γίνεται αυτό. Ε, οπότε έχει αποτελματωθεί συζήτηση. Είχαμε μια τεχνική ανταλλαγή απόψεων για άλλα σημεία, αλλά σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής διαφωνούμε. Αν το λύσουμε αυτό, ε, πολύ γρήγορα θα λυθούν και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Και πάλι υπάρχει προθυμία να επιτυχθεί κάποια ευελιξία. Αυτή τη στιγμή όμως, ε, σας επαναλαμβάνω, είμαστε σε τέλμα. Εγώ χάρηκα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την περίπτωση κινήθηκε και έδειξε να έρχεται πιο κοντά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ενδιαφέρεται για την ποιότητα της νομικής συνδρομής, δηλαδή με κριτήρια βάσει των οποίων μπορεί κάποιος να έχει ε, νομική αρρωγή. Ε, σε κάποιες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνονται αυτά και θέλει να μπουν και στην οδηγία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μέλημα του Κοινοβουλίου. Καλό είναι λοιπόν να έχουμε την Επιτροπή στο πλευρό μας. Το πεδίο εφαρμογή, επαναλαμβάνω, είναι πρόβλημα ε, στο τελευταίο τριμερή διάλογο συμφωνήσαμε τώρα ε, να κοιτάξει το Συμβούλιο να μας πει ποια είναι τα δικά τους προβλήματα. Γιατί δεν δέχονται αυτό που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Δεν ξέρω αν είναι νομικά ε, τα επιχειρήματα ή όχι. Η Προεδρία δεσμεύτηκε να τα συζητήσει αυτά τα θέματα με τα κράτη-μέλη και να φέρουν έγγραφο. Χρειάστηκε μάλλον περισσότερο χρόνο από ότι προβλέπαμε. 20 Οκτωβρίου είναι επόμενη ημερομηνία για το τριμερή διάλογο και μετά από αίτημα της ε, Προεδρίας της Λουξεμβουριανής ε, ματαιώθηκε και η επόμενη συνεδρίαση θα πάει μάλλον τον Νοέμβριο. Καταλαβαίνω ότι θέλει η Προεδρία πριν γίνει η νέα συνάντηση να έχει κάτι χειροπιαστό και ένα συγκεκριμένο έγγραφο και όχι να έρθουμε για τρίτη φορά και να επαναλάβουμε αυτά που ακούσαμε την πρώτη και τη δεύτερη. Τέλος, ε, χαίρομαι πάρα πολύ για τη συνεργασία με τους σκιώδεις ηγητές. Ε, κάθε φορά συνεννοούμαστε πώς ε, θα τοποθετηθούμε. Εμείς τηρούμε την ίδια στάση που είχαμε δεν ακούμε κανένα επιχείρημα, τουλάχιστον εύστοχο ή που να ευσταθεί επιχείρημα από το Συμβούλιο γιατί να αποστούμε από αυτή τη θέση μας. Ας περιμένουμε λοιπόν το έγγραφο και βλέποντας και κάνοντας. Αυτή τη στιγμή δύσκολα τα πράγματα και σκοτεινά. Δεν κινείται καθόλου το Συμβούλιο και θα πρέπει να ξέρουμε ότι μετά την Προεδρία του Λουξεμβούργου ακολουθούν οι κάτω χώρες που ήταν και επιφυλακτικές βέβαια, έτσι και αλλιώς για την οδηγία αυτή και το πεδίο εφαρμογής και το εύρος που θέλει το Κοινοβούλιο. Και μετά έχουμε προεδρίες που δεν ενδιαφέρονται καθόλου σχεδόν, πάρα πολύ. Οπότε θα πρέπει να φροντίσουμε αν θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα να γίνει φέτο, αλλιώ το πρώτο εξάμεινο του 2016 κατά τη διάρκεια τη Ολλανδική Προεδρία. Σταματώ εδώ. Αν έχετε ερωτήσει, με χαρά να τι απαντήσω. Thank you very much, uh, Ευχαριστούμε, κύριε Δεγιόμ. Από τους συναδέλφους πρώτος ο κύριος Μισελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δείχνουμε αποφασιστικότητα ώστε η οδηγία αυτή να προσφέρει υποστηθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρόταση είναι συνεκτική και είναι επιπλέον βήμα πρόοδου για την οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού ποινικού χώρου με την προσωρινή και τακτική δικαστική συνδρομή και με εγγύηση για την ανάκτηση εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών. Επίσης δεν θέλουμε ένα σύστημα δικαιοσύνης δύο ταχυτήτων. Δεν γίνεται όσοι δεν έχουν τα απαραίτητα μέσα να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε έναν συνήγορο ή δικηγόρο από τη στιγμή που τους θερούνται οι ελευθερίες τους. Επίσης, η αμεροληψία δικαιο... της λήψης αποφάσεων από τις δικαιοδοσίες, η ανεξαρτησία των αρχών που λαμβάνουν τις αποφάσεις πρέπει να προασπιστούν, να τις προασπιστούμε μάλλον, ώστε να είναι σαφές ότι λαμβάνουν τις αποφάσεις τους ε, ουδέτερα. Οι προτάσεις αυτές προστατεύουν το δικαίωμα υπεράσπισης και νομικής συνδρομής και δείχνουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι τα δικαιώματα στέρησης της ελευθερίας ή μη στέρησης της ελευθερίας τους είναι κάτι που μας αφορά άμεσα και λαμβάνουμε μέτρα γι' αυτό. Προέδρο. ευχαριστούμε κύριε Μισελ. Ξέχασα να πω ότι θα ισχυωδήσω συγκεκριτής από το φιλελεύθερο για θέμα αυτό, η κυρία Σίπχελ, από του σοσιαλιστέ και Can... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Καταρχά εκτιμώ τη δουλειά του Ντένι και τη συνεργασία του με τις συζητητές, αλλά και όσον αφορά τον τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο. Συμφωνώ μαζί του ότι Χρειαζόμαστε στην έκθεση πιο ευρύες συστάσεις. Στις συζητήσεις με το Συμβούλιο πάντα καταλήγουμε στο ίδιο θέμα, ότι όταν μιλάμε για τα δικαιώματα των πολιτών, μιλάμε για το κόστος, όταν μιλάμε για άλλα θέματα όμως, εξοδεύουμε εκατομμύρια. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σαφείς εδώ. Δεν έχει νόημα να αναφερόμαστε στο δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο, αλλά όποιος δεν μπορεί να πληρώσει τελικά να μην μπορεί να ε, απολαύσει αυτό το δικαίωμα. Για να καταλήξουμε σε συμβιβασμό χρειαζόμαστε σαφή επιχειρήματα από πλευρά του Συμβουλίου και δεν έχουμε καταλάβει γιατί δεν, γιατί δεν μπορούν να μετακινηθούν στις θέσεις τους. Θα εμείνουμε λοιπόν και εμείς στη θέση μας και ελπίζουμε το Συμβούλιο να μας δώσει κάτι πιο συγκεκριμένο σχετικά με το γιατί έχει διαφορετική άποψη, ώστε σε μελλοντικέ συναντήσεις να έχουμε εις βάθος συζητήσεις. Προς το παρόν όμως θα εμείνουμε στη θέση μας εμείς οι σκιώδες εισηγητές. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ντένις, έχετε κάποιες ε, τελευταίες παρατηρήσεις. Ε, πάρα πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Χαίρομαι για την υποστήριξη των σχεδόν εισηγητών και των απόντων σήμερα. Είμαστε πάρα πολύ συμπαγής ομάδα και καλή και ακριβώς και χάρη σε αυτή την ενότητα μπορούμε να ασκήσουμε πίεση στο Συμβούλιο. Βλέποντας και κάνοντας λοιπόν θα περιμένουμε τον Νοέμβριο αν θα προκύψει τίποτα και ελπίζω να είναι καλύτερα τα νέα από τα σημερινά. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε συνάδελφοι στο σημείο 4. Την απόφαση για την υπόθεση του Μαξιμίλιαν Σρέμ στην υπόθεση για τον ασφαλή λιμένα. Θα ακούσουμε εδώ την νομική μας υπηρεσία, η οποία θα παρουσιάσει αυτή τη σημαντική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 6ης Οκτωβρίου 2015 και θα δώσω το λόγο στον κύριο Καγιόλα ή ο κύριος Μουρ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, φαντάζομαι ότι όλοι γνωρίζετε τα πορίσματα αυτή τη υπόθεση ε, πλέον. Στην ε, ανώτατο σχηματισμό του το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν μπορεί να ισχύσει η απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ασφαλή λιμένα. Η οδηγία 9566 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να επιτρέπει πάντοτε στι εθνικέ αρχέ να διερευνούν αυτά τα ζητήματα. Πολύ σύντομα θα δώσω την επισκόπηση των ε, γεγονότων που έχουν να κάνουν με την υπόθεση αυτή και μετά θα σχολιάσω το περιεχόμενο της απόφασης. Τι αφορά λοιπόν αυτή η υπόθεση, οι περισσότεροι το γνωρίζετε, αφορά την μεταφορά προσωπικών δεδομένων από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ της Αμερικής. Ο Μαξ Σρέμς απευθύνθηκε στις Ιρλανδικές Εθνικές Αρχές για να ερευνήσουν την προσφυγή του, δηλαδή τη μεταφορά από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ που θεωρήθηκε μια ασφαλή Μετά τι αποκαλύψεις του Edward Snowden. Η Ιρλανδική Αρχή αρνήθηκε να ερευνήσει το θέμα αυτό, ισχυριζόμενη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αποφασίσει, βάσει τη απόφαση ασφαλού λιμένα, τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων προ τι ΗΠΑ που είναι ασφαλή, διότι υπάρχει επαρκέ επίπεδο προστασία βάσει τη οδηγία. Ο κ. Σρέμ ε, προσέβαλε αυτή την απόφαση στο Ιρλανδικό δικαστικό σύστημα το ζήτημα έφτασε στον Νότο το Δικαστήριο της Ιρλανδίας και ο δικαστής αποφάσισε να παραπέμψει το ερώτημα αυτό προδικαστικό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ιδίως για την ερμηνεία της οδηγίας υπό το φως της χάρτας. Έτσι προέκυψε όλη αυτή η υπόθεση. Απλώς να επισημάνω ότι ο Ιρλανδός δικαστής δεν ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αποφασίσει το κατά πόσο ισχύει και μπορεί να ισχύει η απόφαση ε, ασφαλούς λιμένα. Όμως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επέλεξε να το κάνει και θα εξηγήσω το γιατί. Γιατί κατέληξε σε αυτό το συμπεράσμα το δικαστήριο με δική του πρωτοβουλία. Επίσης, να εξηγήσω γιατί το Ευρωκοινοβούλιο αναμίχθη σε αυτή την υπόθεση. Το Κοινοβούλιο επέβαλε τις παρατηρήσεις του για το θέμα αυτό, όπως ξέρετε πριν από ένα χρόνο περίπου, και η Επιτροπή σας μας στήριξε σε αυτό προκειμένου να διασφαλίσει ότι η οδηγία ερμηνεύεται σωστά βάσει της χάρτας. Τελικώς, το δικαστήριο θεώρησε ότι η οδηγία συνάδει πλήρω με την χάρτα. Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση, η περίπτωση να μην συμφωνούν και να μην συμβαδίζουν. Δεν υπήρχε, λοιπόν καμία αμφισβήτηση προ αυτό από το δικαστήριο και ακριβώ επειδή συμβαδίζει με την χάρτα η οδηγία, η απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κηρυχθεί άκυρη. Διότι το δικαστήριο αποφάσισε ότι αυτό που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συνάδει ούτε με τη χάρτα ούτε με την οδηγία. Μια πολύ γενικόλογη παρατήρηση πρώτα απ' όλα. Είναι προφανέ ότι η υπόθεση αυτή προέκυψε γιατί ακριβώ ένα μεμονωμένο πολίτη αποφάσισε να προσφύγει για το θέμα αυτό. Αν ο Μαξ Σέμ δεν είχε ζητήσει από την Ιρλανδική Αρχή Προστασία των Δεδομένων να ερευνήσει το θέμα αυτό, και αν είχε αρνηθεί η Ιρλανδική Αρχή να το ερευνήσει, δεν θα είχε προσφύγει στα Ιρλανδικά δικαστήρια. Ε, ο κ. Σέμ και η οδηγία Safe Harbor θα ασφαλισμένα θα ίσχυε ακόμα σήμερα κανονικά. Ο Ιρλανδό Δικαστή, που εξέτασε την υπόφαση αποφάσισε να την παραπέμψει, να την αναπέμψει μάλλον στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και ο κύριος Χόγκαν ο δικαστή Χόγκαν δεν ήταν υποχρεωμένο, επέλεξε να το κάνει. Για τα Ιρλανδικά δικαστήρια λοιπόν το θέμα ήταν άκρο σημαντικό προφανώ και έπρεπε να επιληθεί ευθύ αμέσω από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Άρα την αναγνώρισή μα πρέπει να την απευθύνουμε κυρίω στον κύριο Σρέμψ αλλά και στα Ιρλανδικά δικαστήρια που έθεσαν το θέμα αυτό και το ε, έφεραν ε, μπρο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ε, εξού και έχουμε καταλήξει στη σημερινή απόφαση. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ιρλανδική Αρχή Προστασία Δεδομένων δεν προστάτευσαν τα θεμελιώδη δικαιώματα με τι δικέ του δυνάμει. Το δικαστήριο θεώρησε ότι πρέπει να παρέμβει για να προστατεύσει τα δικαιώματα των πολιτών. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε από αυτό το φω τη συγκεκριμένη υπόθεση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δραματίσει εδώ θετικό ρόλο. Ιδίω προωθώντα την άποψη ότι όλοι οι κανόνε της, ε, του ευρωπαϊκού δικαίου, είτε είναι οδηγίε είτε αποφάσει τη Επιτροπή, όλοι οι κανόνε θα πρέπει να ερμηνεύονται βάσει και ε, συμβαδίζοντα με την χάρτα. Αυτό είναι μια παρατήρηση ουσία ε, επί τη απόφαση. Ίσως η πλέον σημαντική. Τώρα για τη συλλογιστική του δικαστηρίου βασίζεται κυρίως στην χάρτα. Και στο πεδίο τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπω καθορίζονται στη Χάρτα, θα πρέπει πάντοτε να γίνονται πλήρω σεβαστά. Όλοι οι κανόνε τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αποφάσει ή οδηγίε, θα πρέπει να ερμηνεύονται βάσει τη Χάρτα. Εάν αυτοί οι κανόνε δεν συμβαδίζουν ή δεν συνάδουν με την Χάρτα, θα πρέπει να λαμβάνει απόφαση αναπερίπτωση το δικαστήριο. Αυτό και συνέβη. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, η οδηγία θεωρήθηκε ότι συνάδει με τη Χάρτα. Το δικαστήριο λοιπόν δεν αφισβητεί σε καμία περίπτωση την ισχύ τη οδηγία. Ωστόσο, το δικαστήριο θεώρησε ότι η απόφαση ασφαλή λιμένα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συνάδει ούτε με τη χάρτα ούτε με την οδηγία, εφόσον ερμηνεύονται σωστά βάσει τη χάρτα. Για τον λόγο λοιπόν αυτό, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κήρυξε άκυρη την απόφαση ασφαλή λιμένα. Αλλά πρέπει να πούμε ότι η χάρτα ε, ισχύει μεν, αλλά προκύπτει το επόμενο ερώτημα. Ερώτημα, ποιο είναι το επίπεδο προστασία που πρέπει να εξασφαλίζεται. Υπ' αυτή την έννοια ήταν σαφέ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι και η χάρτα και η οδηγία ε, απαιτούν υψηλό επίπεδο προστασία. Και αυτό ίσω είναι η σημαντικότερη λέξη, η λέξη κλειδί που πρέπει να ακολουθήσουμε σε όλη την εξέταση τη απόφαση του δικαστηρίου. Υψηλό επίπεδο προστασία. Υψηλό επίπεδο προστασία βέβαια δεν πρέπει να ε, νοείται μόνο σε επίπεδο προστασία εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και να διασφαλίζεται εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, όταν τα δεδομένα μεταφέρονται από την Ευρώπη προ ε, τρίτη χώρα, αυτή η τρίτη χώρα πρέπει να προσφέρει επαρκέ επίπεδο προστασία. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει και εκεί υψηλό επίπεδο. Το δικαστήριο διευκρινίζει ότι οι τρίτε χώρε δεν πρέπει να έχουν πανομοιότυπο επίπεδο προστασία με αυτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει δυνατότητα ευελιξία, μπορούν οι τρίτε χώρε με άλλου τρόπου να αποδεικνύουν ότι προστατεύουν τα δεδομένα, έχουν και άλλα μέσα στη διάθεσή του και υπάρχει και ένα πρόγραμμα πιστοποίηση βάσει τη απόφαση και αυτό που προβλέπουν οι Ηνωμένε Πολιτείε θεωρείται αποδεκτό και αυτό μπορεί να γίνει γενικώ παραδεκτό. Όμω το δικαστήριο θεωρεί ότι το επίπεδο προστασία προκειμένου να είναι ακριβώ υψηλό πρέπει να είναι αντίστοιχο τουλάχιστον από την πλευρά τη τρίτη χώρα. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι το δικαστήριο επιμένει ότι η νομική τάξη, η νομοθεσία τη τρίτη χώρα πρέπει να προβλέπει το υψηλό αυτό επίπεδο προστασία. Πρέπει να υπάρχει χωρή νομοθεσία λοιπόν, οι διεθνεί δεσμεύσει που να δεσμεύουν τι δημόσιε αρχέ τη τρίτη χώρα να σεβαστούν το υψηλό επίπεδο προστασία. Δεν αρκεί οι ιδιωτικέ εταιρείε να αναλαμβάνουν από μόνε του κάποιε υποχρεώσει. Αυτό δεν αρκεί. Και αυτό είναι ένα από του βασικού λόγου που το δικαστήριο τελικώ συμπέρανε ότι η απόφαση του ασφαλώ λιμένα δεν είναι η κατάλληλη ε, για τι περιπτώσει αυτέ. Γι' αυτό ακριβώ το δικαστήριο αποφάσισε να κηρύξει άκυρη την απόφαση ασφαλής λιμένος. Στην πραγματικότητα, ο βασικός λόγος που θεώρησε ότι το δικαστήριο ότι η απόφαση αυτή είναι άκυρη είναι επειδή επειδή βάσει τη οδηγία δεν είναι ακριβώς η κατάλληλη, δεν είναι εύστοχη απόφαση. Μια απόφαση τέτοιου είδους θα πρέπει να εξετάζει την εθνική νομοθεσία μιας τρίτης χώρας και βάσει αυτής να κρίνει αν το επίπεδο προστασίας της είναι υψηλό ή όχι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως την απόφαση της δεν δήλωσε ότι η νομοθεσία των ΗΠΑ, το νομικό του σύστημα προσφέρουν το επαρκέ στο υψηλό επίπεδο προστασίας που απαιτείται. Απλώς υπήρχε ένα σύστημα πιστοποίησης και αυτό δεν είναι αρκετό. Για τον απλούστατο λόγο ότι η απόφαση, και για αυτόν τον απλούστατο λόγο έπρεπε η απόφαση ασφαλής να κηρυχθεί άκυρη. Όμω το δικαστήριο δεν περιορίστηκε σε αυτό το απλό Προχώρησε και περαιτέρω έδωσε κάποιε πολύ σημαντικέ ε, γραμμέ, αδρέ γραμμέ, που θα ισχύουν πλέον για όλε τι ε, υποθέσει. Όπω ε, την όπως κάποιες βασικές αρχές για το πώ θα εφαρμόζονται η χάρτα και η οδηγία. Πρώτα απ' όλα ότι η νομοθεσία δεν μπορεί να επιτρέπει τη μαζική παρακολούθηση στην πράξη. Εδώ δεν μιλάει για την νομοθεσία τρίτων χωρών ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το σημείο αφετηρία είναι η νομοθεσία εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποτέ δεν μπορεί να επιτρέπεται τη μαζική παρακολούθηση. Θα πρέπει να είναι σαφέ. Mass surveillance, μαζική παρακολούθηση, είναι ορολογία που χρησιμοποιώ εγώ. Δεν τη χρησιμοποιήσατε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην διατύπωσή του ο Ιρλανδός Δικαστή, όταν ε, παρέπεψε την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο χρησιμοποίησε παρόμοια διατύπωση, όμω το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν το είπε ακριβώ έτσι. Μίλησε για πρόσβαση σε γενικέ γραμμέ σε όλο το περιεχόμενο τη ηλεκτρονική επικοινωνία. Αυτό ουσιαστικά είναι μαζική παρακολούθηση. Είναι μια ακραία περίπτωση. Εάν λοιπόν δεν είναι δυνατόν εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο κάτω μέλου ή ευρωπαϊκό επίπεδο, να προβλέπει και να επιτρέπει τέτοιε ακραίε μορφέ παρακολούθηση, τότε δεν μπορεί να αποδεχόμαστε μια τρίτη χώρα να κάνει κάτι τέτοιο, εφόσον απαντούμε επαρκέ επίπεδο προστασία. Και εφόσον σε αυτή τη χώρα μπορεί να υπάρχει μαζική παρακολούθηση σε γενικευμένο επίπεδο για τι ηλεκτρονικέ επικοινωνίε. Αυτή η αρχή λοιπόν ε, διατυπώνεται σαφώ, θα παραβιαζόταν η χάρτα λόγω του βασικού δικαιώματο προστασία του ιδιωτικού βίου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό κάτι τέτοιο. Η δεύτερη αρχή που διατυπώνει το δικαστήριο στην απόφασή του έχει να κάνει με το δικαίωμα να προσφύγει κανεί, να ε, καταφύγει σε ένδικα μέσα. Εδώ το δικαστήριο σωστά ε, αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχουν ένδικα μέσα στη διάθεση των πολιτών. Εφόσον οι τέτοιες χώρε δεν το προβλέπουν αυτό, εφόσον ο πολίτης δεν μπορεί να προσφύγει ε, για την ε, προστασία των δικαιωμάτων του ιωτικού βίου ή την προστασία των δεδομένων, δεν μπορεί να θεωρηθεί το επίπεδο προστασία επαρκέ. Για δύο λόγου το δικαστήριο δηλώνει ότι η τρίτη χώρα δεν μπορεί καταρχήν να θεωρηθει το επιπεδο προστασιας επαρκες για δυο λογους το δικαστηριο δηλωνει οτι επίπεδο προστασίας εφόσον η νομοθεσία επιτρέπει την μαζική παρακολούθηση ή είτε ε, ε, υπάρχει απουσία ε, άσκησης ένδικων μέσων για τους Ευρωπαίους πολίτες στην τρίτη χώρα. Οι δύο λοιπόν αυτές αρχές νομίζω ότι θα είναι ιδιαίτερα εύστοχες για υποθέσεις που μπορούν να προκύπτουν στο μέλλον. Το δεύτερο ζήτημα όπου τοποθετείται το δικαστήριο και είναι πολύ σημαντικό είναι το θέμα της ερμηνείας της ισχύουσας οδηγίας. Εδώ το δικαστήριο ήταν πολύ σαφές. Η οδηγία σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περιορίσει τι αρμοδιότητε τη των ε, εθνικών αρχών ε, προστασία των δεδομένων. Σε καμία περίπτωση η Επιτροπή δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Επιβεβαιώνει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ε, το Δικαστήριο με την απόφασή του, δεν δίνουν σε καμία περίπτωση τέτοιε αρμοδιότητε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με την απόφαση όμω του ασφαλού λιμένα, σαφώ περιορίζει τι αρμοδιότητε και τι εξουσίε των Εθνικών Αρχών Προστασία των Δεδομένων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εδώ παρε, ε, υπερβαίνει τι ε, εξουσίε τη. Γι' αυτό λοιπόν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κηρύξε άκυρη την απόφαση ασφαλή λιμένα. Πρέπει να μπορούν οι εθνικές αρχές να διερευνούν τέτοιες προσφυγές, όπως αυτή που εξετάζουμε σήμερα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατέληξε στο πορισμά ότι υπάρχει πρόβλημα με την μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες και θα πρέπει η εθνική αρχή, εφόσον προκύψει πρόβλημα, να μπορεί να επιτρέψει να ε, εξεταστεί η υπόθεση από το Εθνικό Δικαστήριο και εφόσον προκύψει πρόβλημα και υπάρξει παρόμοια κατάσταση όπω η σημερινή, να μπορεί να αναπευθεί η υπόφαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κάτι που ήδη έγινε και η απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κηρύχθηκε άκυρη. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλέ ερωτήσει από του ε, βουλευτέ. Θα σταματήσω εδώ και είμαι στη διάθεσή σα για να απαντήσω σε ερωτήσει. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε για πρώτη φορά θα ρωτήσω την Κομισιόν πώς σκοπεύει να συμμορφωθεί με όλα αυτά και θα ήθελα να πω στην Επιτροπή μας ότι θέλουμε να δούμε την κυρία Ιερόβα και το είπα την προηγούμενη εβδομάδα ότι θέλουμε να την δούμε άμεσα και μάλιστα θέλουμε να μιλήσει στο σύνολο της Επιτροπής και όχι μόνο στους συντονιστές και να μας πει πώς η Κομισιόν θα συμμορφωθεί με την απόφαση. Θα επικεντρωθούμε λοιπόν στο τι θα κάνει η Κομισιόν. Θα ήθελα τώρα να ακούσουμε τους Ευρωβουλευτές, μετά το Συμβούλιο και την Κομισιόν και μετά ε, να ακούσουμε τις απαντήσεις της νομικής υπηρεσίας. Όλοι θα έχουν διαβάσει την απόφαση. Σας παρακαλώ λοιπόν να μας υποβάλλετε τις παρατηρήσεις σας, διότι το Κοινοβούλιο έχει συμμετάσχει σε αυτό το νομικό αλλά και πολιτικό αποτέλεσμα. Για να Άλπρεχτ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, θα ήθελα να συμφωνήσω με την νομική υπηρεσία όσον αφορά τον ρόλο του Max Schrems και την αφοσίωσή του στο θέμα αυτό, ώστε να βγει μια τέτοια απόφαση που αφορά όλους τους καταναλωτές στην ευρωπαϊκή αγορά. Εάν ε, δεν υπήρχε αυτό, ακόμα θα θερούμασταν κάποια θεμελιώδη δικαιώματα, κάτι που ισχύει εδώ και 15 χρόνια. Είναι λοιπόν σημαντικό να τονίσουμε ότι προφανώς κάτι πήγε στραβά εδώ. Διότι εάν το δικαστήριο πρέπει να εκδώσει απόφαση που να θέτει ένα αμφιβόλο το όλο σύστημα του ασφαλούς λιμένα μετά από 15 χρόνια, αυτό δεν δίνει πολύ καλή εικόνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω λοιπόν ότι τώρα εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγνωρίσει ότι κάποια πράγματα στον τομέα αρμοδιοτήτων της πήγαν στραβά. Και αυτό δεν μπορεί να διορθωθεί βιαστικά. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης να αναγνωρίσει ότι το δικαστήριο θεώρησε το νομικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών ανεπαρκές όσον αφορά την επαρκή προστασία υπό το φως αυτής της οδηγίας. Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν τώρα που έχουμε την απόφαση που ο κόσμος ε, λέει «Ωραία, ας ε, έχουμε τότε έναν νέο ασφαλή λιμένα, Safe Harbor Plus». Πώς μπορούμε να αλλάξουμε το νομικό καθεστώς στις Ηνωμένες Πολιτείες με απόφαση του, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει. Τελεία και παύλα. Νομίζω ότι αυτό είναι το μόνο που έχουμε να πούμε σχετικά με την απόφαση. Δεν μπορεί να υπάρξει Safe Harbor Plus, νέο καθεστώς ασφαλούς λιμένα, σε αυτό το νομικό πλαίσιο. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να στείλει ακριβώς το μήνυμα από την πρώτη ημέρα έκταση της απόφασης στους εταίρους μας στις ΗΠΑ ότι θα πρέπει εκείνοι να μας παρουσιάσουν μια ικανοποιητική λύση. Δεν υπάρχει νομική βάση στον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ε, συνθήκη ε, του ΓΕΣ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σχετικά με την προστασία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες να παράσχουν ένα επαρκές καθεστώς για την προστασία δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν υπάρχει άλλο σύστημα παροχής επαρκούς προστασίας σε σχέση με την οδηγία για την προστασία των δεδομένων του 1995. Γνωρίζοντας αυτό, η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ε, ισχνή. Εγώ είμαι απογοητευμένος. Πιστεύω ότι και οι καταναλωτές είναι απογοητευμένοι. Διότι οι καταναλωτές ε, πρέπει να καταναλώνουν χρόνο δικό τους και χρήμα, να προσφύγουν πρώτα σε εθνικό δικαστήριο, να βρουν δικηγόρο. Ε, κατά λάθος λέει ο μιλητής ε, να προσλάβουν δικαστήριο, όχι βέβαια δεν μπορούν να προσλάβουν δικαστήριο, αλλά από ό,τι κατάλαβα είναι αρκετά ε, δαπανηρό στην Ιρλανδία να ε, προσλάβει κανείς δικηγόρο και μετά να προσφύγει ο πολίτης στο δικαστήριο ε, στο Λουξεμβούργο και τελικά να μην λαμβάνεται σοβαρά η απόφαση. Αυτό το μήνυμα θα πρέπει να το αποφύγουμε. Θα πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά την απόφαση αυτή και να δείξουμε ότι αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι κάτι το οποίο υπάρχει στην ε, συνθήκη δεν νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό να ελπίζουμε σε αλλαγή της συνθήκης, ε, ακόμα και αν πιστεύω ότι υπάρχουν άλλα πράγματα στις συνθήκες που θα πρέπει να αλλάξουν. Η Κορνίλια Έρνστ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε θερμά τον ε, αυστριακό φοιτητή Μαξιμίλιαν Σρέμς που ε, τα έβαλε με ένα πρόβλημα το οποίο φαινόταν ότι δεν μπορεί να λυθεί. Έχουμε λοιπόν τώρα νομικές συνέπειες ε, και θα πρέπει να υπάρξουν αντιδράσεις ε, και διαπιστώνουμε ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιες ε, είναι οι νομικές συνέπειες. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι ασφαλή στις ΗΠΑ. Πολιτείες όσο τέλεια και να τα ελέγξουμε όλα, όσο τέλειο και να είναι το σύστημα, πάντα υπάρχει ένα σύστημα. Λόγω της ε, εθνικής ασφαλείας, η, ε, τα προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών πρέπει να διαβιβάζονται. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και έχω την εξή ερώτηση. Ποια είναι εδώ η διέξοδος. Ε, θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια διαφορετική συζήτηση σχετικά με την... Ε, εθνική ασφάλεια. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τέτοια που ποτέ δεν θα είναι ασφαλή τα δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών. Το άλλο θέμα είναι ότι πάει ο ασφαλής λιμένας. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε πολύ αυτό. Η οδηγία αυτή είναι άκυρη. Δεν χρειαζόμαστε μια τέτοια οδηγία. Πρέπει να έχουμε έναν καλό βασικό κανονισμό όπου να θεσπίζονται οι διατάξεις σχετικά με τα ε, προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση. Αναφέρεται η επαρκής προστασία. Για μένα λοιπόν τίθεται το ερώτημα. το DPA πώς μπορεί να το ελέγξει αυτό. Τι, νομική, τι νομικά κανάλια υπάρχουν εδώ ή μήπως χρειαζόμαστε και εδώ έναν Max Schrems. Τι συνέπειες θα υπάρξουν σε άλλες συμφωνίες και συμβάσεις. Ευχαριστώ, η Σοφία Νετφέλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Την τελευταία εβδομάδα Είδα πολλές αντιδράσεις θυμού, πανικού και αγανάκτησης ως προ την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αλλά αυτό που έκανε το δικαστήριο είναι να ε, αποτιμήσει τον νόμο ε, όσο και αν ε, αυτό ευνηδίασε σε κάποιους ε, ακόμη και αν ήταν η πρώτη υπόθεση που αφορούσε το Safe Harbor καλά έκανε διότι η απόφαση ασφαλώς λιμένα από η σειρά ετών είχε αφισβητηθεί μπορεί λοιπόν να αποτελεί αυτό έκπληξη αλλά το επιχείρημα ότι χρειαζόμαστε χρόνο για να δούμε όλες τις συνέπειες μέσα της απόφασης είναι επίσης σωστό. Απλώς θα ήθελα να ξέρω λίγα περισσότερα για τις επιπτώσεις. Η ομάδα μου, η ομάδα ALD, έχει γράψει στους επιτρόπους Timmermans, ε, Γιούροβα και Αβραμόπουλο για να δούμε ακριβώς αυτή η συμφωνία ή η συμφωνια DFTP, ε, η συμφωνία Ομπρέλα, η συμφωνία για την ε, η εισαγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποφάσεις για υπηρεσίες πληροφορικές που δεν βασίζονται στις ευρωπαϊκές, ε, στα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και επιχειρηματολογία για εθνικούς νόμους για τη μαζική παρακολούθηση, όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Διότι υπάρχουν τουλάχιστον τρία παραδείγματα των μελών, όπου δεν είναι καθόλου ούτε καν κοντά στην επίτευξη των προτύπων που θέτει το δικαστήριο τα άλλα εργαλεία που ανέφερε την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αντί του ασφαλού λιμένα, όχι, δεν συμφωνώ, γιατί αν μπορούσαν να αποκαταστήσουν τον ασφαλή λιμένα, θα γινόταν αυτό τα τελευταία 15 χρόνια. Άρα, δεν είναι αυτή η εναλλακτική. Πρώτα λοιπόν πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες ε, συνολικά και μετά να δούμε τι θα πρέπει να κάνουμε εμείς. Χρειάζεται μια νέα διαθέτηση. Δεν ξέρω πώ θα την ονομάσουμε. Safe Harbor Sin, ε, κάτι άλλο. Αλλά το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητέ. Υπάρχει ένα βασικό στοιχείο εδώ. Ότι οι αρχές των ΗΠΑ πρέπει να κινηθούν. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι πάντοτε τις διακλαδικές μας σχέσεις τις αντιμετωπίζουμε με διαφορετικά μέτρα και σταθμά από ό,τι με τις άλλες χώρες. Εντάξει, γίνεται για πολιτικούς λόγους αυτού, αυτό, κάποιες φορές είναι δικαιολογημένο, αλλά δεν είναι αυτό επιχείρημα για τον οποιοδήποτε δικαστή. Θα πρέπει να δει μόνο το κατά πόσο να ευσταθεί νομικός ε, ο δικαστής σε κάθε περίπτωση. Άρα ε, το να εφαρμόσουμε τους κανόνες του δικαστηρίου δεν είναι θέμα του αν μας αρέσει ή όχι, πρέπει να το κάνουμε θέλουμε δεν θέλουμε. Άρα πρέπει να συνεχίσουμε με, να μεταφέρουμε δεδομένα ε, από την άλλη όχθη του Ατλαντικού. Εντάξει, το θέλουμε αυτό. Δεν θέλουμε να οριοθετήσουμε το διαδίκτυο, το ίντερνετ, ούτε να έχουμε προστατευτισμό, ούτε να αποκόψουμε του εαυτού μα από όλα τα ωφέλη τη ανοιχτή οικονομία και του ανοιχτού ίντερνετ. Όμω θα πρέπει και οι ΗΠΑ από την πλευρά του να δείξουν ότι και αυτέ τι ενδιαφέρει. Θα πρέπει να κινηθούν. Λέμε ότι έχουμε κοινά πρότυπα. Εφόσον έχουμε λοιπόν κοινέ αξίε, α φροντίσουμε να το δείξουμε αυτό λίγο στην πράξη. Ένα τρίτο θέμα, ε, και τελευταίο πρόεδρε, είναι ότι εδώ δεν είναι μόνο ένα ζήτημα μια μονομένη δικαστική απόφαση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Είναι θέμα διακυβέρνηση και ποιότητα τη ε, θέσπιση νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να έχει καλύτερη νομοθεσία όπω επαγγελίζεται, αλλά για την ώρα αυτό δεν ισχύει. Είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο. Διότι ο ασφαλή λιμένα το ήξεραν όλοι είχε ένα σωρό ελαττώματα. Δεν ε, θεωρήθηκε άκυρος από το δικαστή την περασμένη εβδομάδα απλώς, αλλά είχε θεωρηθεί ε, εδώ και πολύ καιρό. Το είχε ζητήσει επανειλημμένο στο Κοινοβούλιο να θεωρηθεί άκυρη απόφαση αυτή. Το ίδιο και για την προστασία των δεδομένων. Ήταν πολύ κακή νομοθεσία αυτή. Και για πολλού από εμά, ε, ιδίω η ομάδα μου που είχε καταψηφίσει τότε, θεωρούσε ότι είναι κακή νομοθεσία. Ότι δεν θα αντέξει στι δοκιμέ. Και σε κάποιε άλλε περιπτώσει είδαμε κακή νομοθεσία να περνάει. Και κακή ε, επιβολή τη. Το σκάνδαλο τη Volkswagen. Η FIFA ίσω είναι μια λίγο διαφορετική περίπτωση, άλλη τάξη μεγέθους, αλλά και πάλι έχει να κάνει με τη σωστή εφαρμογή των κανόνων. Έχουμε λοιπόν κάποιου κανόνε για τη διαπτωρεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα γίνει, δεν ισχύει για την ε, FIFA ή το σύστημα αυτό ε, και θα λαμβάνονται αποφάσει αλλού. Εδώ λοιπόν Πρέπει το ζήτημα να το δούμε λιγάκι και υπό το πρίσμα της ποιότητας της, ε, του σχεδιασμού νομοθεσίας, του πώς ε, η νομοθεσία αυτή υλοποιείται και της όλης μας διακυβέρνησης. Και να ολοκληρώσω λέγοντας ότι δεν μπορούμε πρόεδρε να αφήνουμε ένας μόνο τολμηρός ισχυρογνώμων και απομονωμένος πολίτης όμως να αμφισβητεί όλο το σύστημα. Σε αυτό το σώμα έχουμε πολλές φορές επικρίνει όχι μόνο το Συμβούλιο και την Επιτροπή, αλλά πρέπει και εμείς οι ίδιοι να κοιτάξουμε τι νομοθεσία εγκρίνουμε. Έχουμε την υποχρέωση νομοθεσία που περνάμε να είναι ε, πραγματικά διάτητη. Και εδώ αυτό θα πρέπει να διασφαλίσουμε. Ευχαριστώ. Γενικά ε, βέβαια θα πρέπει να κοιτάμε και το χρόνο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η απόφαση και θέλετε να ε, πείτε τη γνώμη σας. Ε, αυτό που είπε η κυρία Βέλτ και άλλοι, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γενικά. Στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα το Σώμα των Επιτρόπων απαντούσε στις Επιτροπές όλη η Επιτροπή και ξέρετε ότι εμείς είμαστε Επιτροπή που ε, φορά ιδιαίτερα το θέμα αυτό και πολλούς επιτρόπους γιατί ε, είναι οριζόντιο έτσι εγκάρσια. Δεν είναι μόνο η κυρία Γιούροβα και άλλοι Επίτροποι. Ο κύριος Άνσιπ μεταξύ άλλων. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θέλουμε να τους δούμε για να εκφράσουμε αυτές τις ανησυχίες μας και θέλω να το ξέρετε. Θέλουμε μεγάλη έτσι, μαζική απάντηση εδώ στην Επιτροπή μας. Η κυρία Λόριστην που είναι και η για την οδηγία έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να συμφωνήσω όμως εκείνους που είπαν ότι ε, κάποιοι ε, ε, ή ένας θαραλέος πολίτης και ε, πείσμων οδήγησε σε επανάσταση στην οτροπία. Το είπε και ε, η Σοφή για τους Αμερικανούς. Είχαμε ένα ε, ε, ε, ανέκδοτο που συναντιέται ένας Αμερικανός με έναν Ρώσο και λέει Αμερικανός είμαστε ελεύθερη χώρα, εμείς μπορούμε να επικρίνουμε τον Αμερικανό Πρόεδρο κάθε μέρα. Λέει και ο Ρώσος και εμείς είμαστε ελεύθερη χώρα και εμείς μπορούμε να επικρίνουμε τον Αμερικανό Πρόεδρο κάθε μέρα. Λοιπόν, ε, κοιτάμε λίγο και τη δική μας αυλή, την προστασία των δεδομένων, όλα τα θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, τι ενδιαφέρει τις επιχειρήσεις και τι ενδιαφέρει την εθνική ασφάλεια. Αυτά τα πράγματα είναι ένα τρίγωνο και ε, λειτουργούν όχι μεταξύ κρατών μόνο, αλλά και εντός των κρατών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το μήνυμα που έστειλε το δικαστήριο και θα πρέπει να κοιτάμε αυτά τα πράγματα με τρόπο πολύ πιο σφαιρικό και ολοκληρωμένο. Από την άλλη, να ξέρουμε και τι γίνεται σε αυτή την ψηφιακή εποχή αναδύεται η Κίνα και η Ρωσία πλέον και ως πάροχη τέτοιων υπηρεσιών. Εκεί να δείτε τι γίνεται και ποια είναι τα προβλήματα πολύ πιο σοβαρά και θα πρέπει να είμαστε πρόθυμοι και έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε και να μην κάνουμε τα στραβά μάτια. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία και πρέπει να πούμε ότι μάλλον αρχίζει μια επανάσταση στις νοοτροπίες και στα μυαλά ε, για τη σημασία και τα γεγονότα και τις επιπτώσεις που έχει αυτή η προστασία δεδομένα. Ευχαριστώ κύριος Μπόνη. Uh, I speak in Polish. I'm sorry. Θα μιλήσω πολωνικά. Κατά τη γνώμη μου, η απόφαση του δικαστηρίου θα πρέπει να θεωρηθεί καταλητική. Χάρη στην απόφαση αυτή, θα αναζητήσουμε μια καλή λύση θα πρέπει να ζητήσουμε αντίστοιχη προσέγγιση από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Και το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν έχουν να κάνουν κάποια πράγματα. Η Κομισιόν διεξάγει συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με ε, τον ασφαλή λιμένα και με τη Γενική Συμφωνία. Εναπόκειται λοιπόν στους Αμερικανούς να επιλύσουν το παρόν πρόβλημα. ευχηθώ τον Γιάννη. Θυμάμαι ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας ε, στη Ουάσιγκτον επισημάναμε την ανάγκη να αλλάξει η νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά ε, τις αρχές περί ιδιωτικού βίου. Ίσως λοιπόν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στείλει μια ευγενική επιστολή στις Ηνωμένε Πολιτείε που να μεταφέρει το σαφές μήνυμα ότι θα πρέπει να κάνουν κάτι για να λύσουν το πρόβλημα. Επιπλέον, η διαβίβαση δεδομένων γίνεται σύμφωνα με κάποιες προϋποθέσεις. αυξάνεται ο ρόλος των ε, εθνικών ε, εποπτών προστασίας δεδομένων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αφήσουμε και από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων να αναθεωρήσει, να εξετάσει τα καθήκοντα των εθνικών ε, επόπτων προστασίας δεδομένων, διότι σε κάποιες περιπτώσεις οι επόπτες έχουν πολλές αρμοδιότητες. Ε, σε άλλες χώρες η κατάσταση δεν είναι εξίσου καλή. Θα ήθελα επίσης κατά την διάρκεια του τριμερούς διαλόγου να αναρωτηθούμε εάν το παρόν σχέδιο πληρεί τις προϋποθέσεις δεδομένου ότι δεν υπάρχει πια η οδηγία για, του, για τον ασφαλή λιμένα. Θα πρέπει λοιπόν το Συμβούλιο να καταλήξει σε σωστή λύση. Η κυρία Σπινέλη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ εξεπλάγιν. Εξεπλάγιν με την έκπληξη των άλλων σε σχέση με την απόφαση αυτή. Γιατί πραγματικά, σε ό,τι αφορά την επανάσταση που έχει να κάνει και με τα ψηφιακά δικαιώματα στην Ιταλία, λόγου χάρη, το συζητάμε εδώ και 15 χρόνια. Και πρόσφατα καταλήξαμε σε μια χάρτα που καταρτίζει και κατοχυρώνει τα ψηφιακά δικαιώματα. Αυτό ε, που ε, φαίνεται είναι ότι τελικά χάρη στη δράση κάποιων πολιτών μας σώζουν οι δικαστές. Χάρη στη δράση κάποιων των μοιρών πολιτών, γιατί είχαμε, έχουμε τώρα τον ε, κύριο Σρέμς, αλλά προηγουμένως είχαμε και τον κύριο Σνόντεν. Μας σώζουν λοιπόν από την αδράνειά μας και ουσιαστικά μεταφράζουν σε πράξη την ε, χάρτα. Ε, δεν αρκεί μόνο η καλύτερη νομοθεσία, αλλά ένα, ένα σύστημα δικαίου που να λειτουργεί στην Ευρώπη. Οι δικαστές λοιπόν και ο ΣΡΕΜΣ μας λένε ότι τα δεδομένα δεν προστατεύονται. Ούτε είναι ασφαλή στις Ηνωμένε Πολιτείες. Πιστεύω λοιπόν και εγώ ότι μπορούμε να μιλήσουμε για μια πραγματική επανάσταση με την απόφαση αυτή, γιατί πραγματικά έρχεται μετά από μια σειρά επεισοδίων και μια, ε, τουλάχιστον μετά από άλλε δύο αποφάσει που αφορούν παρομοίω την προστασία των δεδομένων, το δικαίωμα στη λύθη του 2014 και από κοινού επιτέλους επιτρέπουν μια επανάσταση που μπορεί να γίνει και στις διάφορες διαπραγματεύσεις με την ακύρωση της απόφασης ε, Safe Harbor αλλά και για το Μητρό Επιβατών και για την ε, Συμφωνία για τις Υπηρεσίες TISA και για την Διατλαντική Συμφωνία TTIP Πρέπει όλα αυτά να επηρεαστούν και να έχουμε και μια δήλωση για τα ψηφιακά δικαιώματα κάποια στιγμή. Όταν αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλω να υπογραμμίσω δύο σημεία τα οποία ε, φάνηκαν εύγλωτα και από την απόφαση. Πρώτον, οι, απόφα, οι αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούν να περιορίζουν τι έρευνε και τι δράσει των εθνικών αρχών. Δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να περιορίζει την εξουσία των εθνικών αρχών. Και αυτό το λέω γιατί συχνά στα κράτη υπάρχουν πρακτικές προστασίας των δεδομένων ε, πιο προηγμένες. Δεύτερη παρατήρηση, οι κρατικές επιχειρήσεις της ε, Αμερικής που είναι εκτός της συμφωνίας παρολυμένα λιμένα ε, και η όλη αυτή, όλος αυτός ο επενιγμός. Εφόσον είναι εκτός της ασφαλώς είναι εκτός και αυτής της απόφασης. Δηλαδή οι υποχρεώσεις αυτές που προβλέπονται από τη συγκεκριμένη απόφαση δεν τις αφορούν είναι ελεύθερες να αδιαφορήσουν για αυτές τις αρχές που προγραμμίζει ακριβώς η απόφαση. Ιδίως εάν θεωρούν ότι συνεισφέρουν στη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Δηλαδή μπορούν να συλλέγουν δεδομένα όπω θέλουν. Τρίτον, η συνεργασία μεταξύ Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να ευχαριστήσω εδώ τον πρόεδρο που φρόντισε να ενημερωθούμε εξωδικά και στο ότι ελπί και με συγκεκριμένα βήματα θα έχουμε καλύτερη συνεργασία στο μέλλον με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι είναι πολλά τα κενά της επικοινωνίας του Κοινοβουλίου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ευχαριστώ τον Πρόεδρο που ε, όλη αυτή τη χρονιά επέμεινε ιδιαιτέρως ακριβώς το πόσο πρέπει να είναι εποφελής η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σπινέλη. Πολύ ευγενικά το είπατε. Είναι ένα θέμα ε, για την Επιτροπή θα επανέλθω στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Μπέρκη Τσίπελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Πρώτον, εκτιμώ πάρα πολύ και χαίρομαι για την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά ταυτόχρονα αυτό γεννάει πολλά ερωτηματικά. Το πρώτο είναι, γιατί στο καλό χρειάστηκε, για να μην πω τίποτα άλλο, να πάει ο Μαξ Ρίμ σε Ιρλανδικό δικαστήριο για να δεήσει επιτέλους το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να πάρει τέτοια απόφαση. Γιατί στο καλό χρειάστηκε όλο αυτό. Εδώ και χρόνια λέμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ασφαλής λιμένας δεν είναι ασφαλής για δεδομένα, δεν είναι ασφαλής για την ιδιωτική ζωή. Και οι πολίτες ρώτησαν εμένα, γιατί δεν προσέφυγες εσύ στο δικαστήριο. Μα εμείς ως κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να εργαζόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Κάθε φορά που υπάρχουν ανησυχία, εμείς να προσφεύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργάζεται μαζί μας και να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις δικές μας ανησυχίες. Θα μπορούσε να είχε εκδοθεί λοιπόν τέτοια απόφαση εδώ και χρόνια. Και κάπως πώς να το πω, έχω ενοχληθεί και συγχυστεί ε, ότι αυτό δεν συμβαίνει μόνο στι Ηνωμένε Πολιτείε, όχι μόνο επειδή δεν παίρνουν σοβαρά υπόψη την ιδιωτική ζωή, αλλά απλή, ε, και μόνο η αναφορά τη έννοια, εθνική ασφάλεια χρησιμοποιείται ω γενική πρόφαση και αόριστη για να κάνει ο καθένα ό,τι θέλει με όλα τα δεδομένα. Αυτό το βλέπουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, συμβαίνει και χρειάζεται αντιμετώπιση. Πολλά λοιπόν είναι τα ερωτηματικά. Πρώτον, τι σημαίνει αυτό για τον ασφαλή λιμένα και για την ανταλλαγή δεδομένων. Τι επιρροή μπορεί να έχουμε εμείς και να ασκήσουμε πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες να αλλάξουν τη νομική τους βάση και τι έλεγχο έχουμε. Αναλαμβάνονται σοβαρά οι επιστοποιήσεις και αν είναι ασφαλή τα δεδομένα. Επίσης τι σημαίνει αυτό για άλλες συμφωνίες που έχουμε με τις Ηνωμένες και πολύ γενικά πώς μπορούμε εμείς να εξασφαλίσουμε ότι με την κείμενη αλλά και τη μελλοντική νομοθεσία θα είμαστε εξασφαλισμένοι και όχι μόνο το Κοινοβούλιο αλλά και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και θα τον ακολουθούν για να μην φτάνουν οι νόμοι στα δικαστήρια αλλά εμείς και τα θεσμικά όργανα να νομοθετούμε με σωστό τρόπο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βάιντεν Χέλσερ. Joseph Βάιντεν Joseph Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ χαίρομαι πολύ που υπάρχει δικαστήριο το οποίο τηρεί το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και μπορώ να, ακόμα να θυμηθώ ότι υπήρχαν κάποιοι που αμφέβαλαν για το κατά πόσο θα είχε σημασία το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ιδού λοιπόν η σημασία του. Και βέβαια μπορεί να είναι και μεγάλη. Και χαίρομαι που το κατάφερε ένας πολίτης, πόσο μάλλον και συμπατριώτης μου, που προσέφηκε στο δικαστήριο. Και Είναι πραγματικά μια ρηξικέλευτη ε, απόφαση. Όταν ένα δικαστήριο αποφαίνεται, ε, τότε αυτό είναι δίκαιο, είναι ε, ε, κάτι που πρέπει κάποιος να δεχτεί και να εφαρμόζει το δίκαιο αυτό. Προσπαθούν κάποιοι να επικρίνουν αυτή την απόφαση και να την αποδυναμώσουν ή να την βραχικυκλώσουν. Είναι μια απόφαση πάρα πολύ σημαντική, ουσιαστική που κλονίζει πολλά. Συζητούμε για ε, την καλύτερη ρύθμιση, το better regulation, μήπως να συζητήσουμε και το better law making, πώς να νομοθετούμε καλύτερα. Για να μην έχουμε τέτοιους κραδασμούς. Τώρα, θα ε, όσα μας αφορούν εδώ στην Ευρώπη μπορούμε μόνοι μας να τα διαμορφώσουμε και να μην προσπαθήσουμε τώρα με ολιγορίες και χρονοτριβές να ε, αναβάλουμε την ε, δράση μας, να πάρουμε αποφάσεις μάλιστα θαραλές, χωρίς αναβολές και παραπομπές σε καλένδες. Γιατί φοβάμαι ότι κάτι τέτοιο κινδυνεύει να συμβεί αν δω τις αντιδράσεις. Πρέπει να εξηγενθεί αυτή η κατάσταση γρήγορα. Και εμείς ως Επιτροπή που είχαμε ανέκαθεν άλλη άποψη, φέρουμε τεράστια ευθύνη να ασκήσουμε αυτή την απαραίτητη πίεση για να λυθούν ε, τα πράγματα με σαφήνεια. Και θα ήθελα να ρωτήσω πώς εκτιμά ο Πρόεδρος και το χρονικό ορίζοντα και το χρονοδιάγραμμα. Πότε μπορούμε να υπολογίζουμε δηλαδή τους επόμενους μήνες να έχουμε τελειώσει. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ ε, είναι σύμπτωση ότι τελειώνουμε με έναν Αυστριακό. Θα ακούσουμε τώρα το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ακούσουμε τον κύριο Μούρ στο τέλος. Ε, έχουμε ε, ξεπεράσει λίγο το χρόνο που είχαμε προβλέψει για το θέμα αυτό, αλλά αυτό είναι απόλυτα κατανοητό δεδομένη τη σημασία του. Τον κύριο Κάρλι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ακούσουμε πρώτα. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως αναφέρατε, η Επίτροπος Σιούρεβα θα συμμετάσχει σε ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σας στις 26 Οκτωβρίου. Πιστεύω. Θα ήθελα να τονίσω ότι όπως ήδη αναφέρθηκε η απόφαση ΣΡΕΜΣ είναι μια σαφής δήλωση για τη σημασία της προστασίας των δεδομένων ως το δικαίωμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωση, συμπεριλαμβανομένου εντός του πλαισίου των ε, διεθνών ε, μεταφορών, διεθνών συμφωνιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητεί πιο ισχυρούς κανόνες, ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την ε, διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες είδαμε ότι όσον αφορά την επιβολή του νόμου έχουμε πετύχει σημαντικά αποτελέσματα χάρη στην βοήθεια και υποστήριξη του Κοινοβουλίου σας. Ε, έχουμε πετύχει αποτελέσματα και όσον αφορά την διαβίβαση δεδομένων ε, για εμπορικούς σκοπούς. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να πετύχουμε ασφαλή ρύθμιση για την ε, διαβίβαση ε, δεδομένων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία της απόφασης του δικαστηρίου. Στο μεταξύ, πιο, πιο βραχυπρόθεσμα, οι προτεραιότητες μας ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η προστασία των δεδομένων που διαβιβάζονται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ε, σαφήνεια σχετικά με το πώς πραγματοποιούνται οι διαβιβάσεις αυτές ε, με τα απαραίτητα εχέγγυα και η σωστή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στην εσωτερική αγορά. Έχουμε ξεκινήσει τις εργασίες μας ε, και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στένα με τις Εθνικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων. Για να διασφαλίσουμε την ενιαία εφαρμογή της απόφασης, για να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό και για να διασφαλίσουμε την ε, σωστή διαβίβαση δεδομένων ε, με τα απαραίτητα εχέγγυα. Η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 η ολομέλεια της ομάδας εργασίας αυτής ε, θα συνεδριάσει ετούτη την εβδομάδα και αυτό θα αποτελέσει σημαντικό βήμα στην άμεση αντίδρασή μας ε, στην ε, νέα αυτή απόφαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Υπάρχει διαδικαστικό. Παρακαλώ να είστε σύντομοι, πολύ σύντομα, διότι με εκπλήσει αυτό που άκουσα, διότι αποτελεί σύνοψη αυτών που ακούμε τις τελευταίες δύο, τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει την, από την προηγούμενη εβδομάδα. Εάν έχω ενημερωθεί σωστά, η Κομισιόν ήθελε να υποβάλει νέο καθεστώς ασφαλούς λιμένα με βάση 13 ε, σημεία που έχει εντοπίσει. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να ελέγξει εάν η επίτευξη αυτών των 13 στόχων θα πετύχει το επίπεδο που υπαγορεύει η απόφαση του δικαστηρίου. Δεν θέλω να ακούσω αυτά που λέτε τα τελευταία δύο χρόνια, αυτά τα γνωρίζω. Θέλω να ξέρω τι έχει αλλάξει έκτοτε και νιώθω αγανάκτηση, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα έπρεπε να έχει μάθει από την ε, απόφαση αυτή ότι δεν βρίσκεται στο σωστό δρόμο και ότι θα πρέπει να αλλάξει στρατηγική. Πρόεδρος. Νομίζω ότι ήταν ε, σημαντικό αυτό που είπατε και θα ήθελα να πω ότι Ε, διαφωνώ με αυτά που είπε η Σόφη, διότι κάποιε συζητήσει δεν τι έχουμε ακούσει, διότι έχουν γίνει και κλεισμένων των ε, θυρών. Δεν έχουμε ακούσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια ακριβώ είναι η στρατηγική και το λέω αυτό διότι ο κύριο Άλπρεχτ πολύ σωστά είπε, και επιτρέψτε μου να το πω αυτό, ότι δεν μπορούμε να έχουμε ε, ασφαλή λιμένα νούμερο 2 ε, και δεν έχουμε ακούσει τις συζητήσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει λοιπόν να τα ακούσουμε από αυτά από την Επίτροπο. Χρειαζόμαστε λοιπόν πολιτική στρατηγική. Θα πρέπει να δούμε τι πολιτικά μηνύματα θα στείλετε στη Γερουσία και στους, ε, στην, ε, στις Ηνωμένες Όπως είπε και ο κύριος Άλπρεχτ. Δεν ξέρω εάν έχετε να προσθέσετε κάτι εδώ ή εάν θέλουμε να περιμένουμε να έρθει η Επίτροπος. Αλλά θα σας δώσω το λόγο να πείτε λίγα πράγματα ακόμα και μετά ε, θα τα αφήσουμε όλα στην Επίτροπη. Παρακαλώ. Δεν έχω πολλά να προσθέσω σε αυτή τη φάση. Απλώς η σύσταση που αναφέρατε, η 13η σύσταση, ε, δίνει έμφαση σε κάποια στοιχεία της απόφασης αυτής. Ξέρετε ότι στην 13η ε, σύσταση αναφέρονται τα θέματα της ε, εθνικής πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Ε, ήδη είναι ένα σημαντικό στοιχείο και ξέρετε ότι προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διευκρινίσουμε το σωστό πλαίσιο. Πρόεδρος. Να ακούσουμε το Συμβούλιο, γιατί με την Επιτροπή θα το ξαναπούμε στις 26 του μήνα. Θα έχουμε και τότε και το χρόνο. Ας ακούσουμε λοιπόν το Συμβούλιο. Η κυρία Βάγκνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα από πλευράς Προεδρίας να, επιση... να πω ότι το Συμβούλιο παίρνει πολύ σοβαρά αυτή την απόφαση, διότι στόχος της Προεδρίας είναι το πρόγραμμα των, ε, του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνη ήταν μάλλον να έχουμε μια προκαταρτική αποτίμηση της απόφασης αυτής. Ε, στις 8 Οκτωβρίου στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνη λοιπόν και θα πρέπει να δούμε και την ολοκλήρωση τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων ω το τέλο τη χρονιά μα. Φαίνεται και επίγον και σημαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Α ακούσουμε και πάλι την νομική μα υπηρεσία για να απαντήσει ενδεχομένω στις παρατηρήσει των συναδέλφων. Κύριε Μουρ, ευχαριστώ και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτικό. διότι η απόφαση βγήκε πριν από λίγε μέρε μόλι και σε αυτή τη φάση απλώς την εξετάζουμε προσεκτικά ω προ όλα τα στοιχεία του περιεχομένου τη. Βεβαίω θα συνδράμουμε την Επιτροπή σας τι ερχόμενε εβδομάδε και μήνε, όπως ακριβώς χρειαστεί, για να δούμε πώς μπορούμε να αποτιμήσουμε μαζί την απόφαση αυτή και να παρακολουθήσουμε πώς ε, θα έχει συνέπειε στην πράξη. Με όλη την προσοχή που τη αρμόζει. Το μόνο που προσθέσω είναι ότι στην συνεδρίαση του Σώματος των Επιτροπών την περασμένη εβδομάδα νομίζω ότι σωστά ακούστηκε το μήνυμα από αυτή την Επιτροπή μας ότι πρέπει οι κανόνες προστασίας των δεδομένων να βασιστούν σε άλλη νομική βάση. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε τους ανθρώπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίοι αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, όχι για την Google και την Amazon α πούμε, αλλά είναι ένα σημαντικό θέμα για την Επιτροπή μας. Εάν όλα πάνε καλά, θα συζητήσουμε με την Επιτροπή στις 26 Οκτωβρίου, αλλά ε, είμαι ανοιχτό σε προτάσεις για να δούμε τι συνέχεια θα έχει το θέμα με όλη την καταπήγουσα σημασία που του πρέπει. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι για την αδελφία τη συζήτηση που είχαμε σήμερα και ευχαριστώ για την Επιτροπή και την νομική μας υπηρεσία. Ευχαριστώ κύριε Μουρ. Τώρα συνάδελφοι να περάσουμε στο επόμενο σημείο, που είναι το σημείο 5 συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διαπραγματεύσεις της ε, Συμφωνίας για τις, για τις εμπορικές συναλλαγές της υπηρεσίας της. Ο κύριος Άλμπρεκτ είναι συγκεκριτής από τον πλευρά της Επιτροπής μας. Γιάνν, έχεις το λόγο. Thank you very much, <clears throat> dear colleague. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι μια γνωμοδότηση για το ψήφισμα της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ως προς τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία ΤΙΣΑ, που είναι η Συμφωνία για τις Εναλλαγές στο τομέα των υπηρεσιών. Και μπέρδεψα με το TTIP, ε, διότι κάνουμε και γι' αυτό γνωμοδότηση, για δύο θέματα κυρίως. Και στην Επιτροπή ΙΝΤΑ λοιπόν εμείς γνωμοδοτούμε για το TTIP ε, και είναι οριζόντια ρήτρα θεμελιωδών δικαιωμάτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό αφορά και τις άλλες συμφωνίες και ήταν μια πάγια δική μας απέτηση για όλες τις συμφωνίες. Εξαίρεση το καθεστώς του ΠΟΕ για την προστασία προσωπικών δεδομένων, άρθρο 14 της Συμφωνίας ΓΚΑΤΣ Εκεί ορίζεται ότι η προστασία προσωπικών δεδομένων και οι αντίστοιχοι νόμοι δεν μπορούν να θεωρηθούν εμπορικός φραγμός σε αυτού του είδους συμφωνίες. Και εμείς επιμένουμε σε αυτό και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται με τέτοιο τρόπο και με τέτοια διατύπωση πάντα μία ρήτρα ε, στη Συμφωνία ΤΙΖΑ. Το σχέδιο γνωμοδότησης που έχω καταθέσει επαναλαμβάνει αυτό που είχαμε πει και στην ε, γνωμοδότησή μας για το TTIP με εξαίρεση φυσικά τις ρυθμίσεις που αφορούν μόνο την επενδυτική συμφωνία και όχι τη συμφωνία της. Όλα αυτά τα θέματα φυσικά δεν τα συζητάμε μόνο διμερώς, αλλά με πολλούς άλλους εταίρους, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ, αλλά και πολλές άλλες τρίτες χώρες Οπότε θα πρότεινα να εγκριθεί σύντομα αυτή η γνωμοδότηση με τις ε, παρατηρήσεις που σας ε, κάνω. Και να είναι και πολύ σφιχτό το χρονοδιάγραμμα για τις τροπολογίες καθώς επίσης και η ψηφοφορία για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε και με το ψήφισμα στην Επιτροπή που είναι η αρμόδια Διεθνού Εμπορίου με εισηγήτρια την κυρία Βιβιάν Ρέντινγκ. Αυτά τα ολίγα πλην μεστά. Με χαρά βέβαια να απαντήσω και στις ερωτήσεις. Thank you, Jan. So the deadline for table... Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 19 Οκτωβρίου. Έγκριση του σχεδίου μου 16 Νοεμβρίου. Να δούμε τώρα από τους κοιόδεις ποιους έχουμε εδώ. Ο κύριος Μισελ για τους φιλελεύθερους. Πολύ γρήγορα, Πρόεδρε. Λόγω τη σημασία τη επικείμενη συμφωνία, είναι ουσιαστική σημασία να τοποθετηθεί το Κοινοβούλιο προκειμένου να δώσει τη σωστή κατεύθυνση στις τρέχουσες διαπραγματεύσει. Θα πρέπει να θέσουμε κάποια ορόσημα ώστε η τελική συμφωνία να ανταποκρίνεται στι προσδοκίε μα. Ευχαριστούμε τον εισηγητή, τον κύριο Άλμπρεχτ, για το εξαιρετικό σχέδιο ομοδότηση και συμπεριλαμβάνει τα βασικά σημεία που είναι σημαντικά και για μα. Πιστεύω ότι μπορούμε να εμπλουτίσουμε με τι εξή παρατηρήσει. Πρώτα απ' όλα, επειδή οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι μέρο ε, των διαπραγματευόμενων πλευρών στη συμφωνία ΤΙΣΑ, έστοχο ε, θα ήταν να μιλήσουμε για την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που κήρυξε άκυρη την απόφαση ασφαλώ λιμένα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την μεταφορά προστασία προσωπικών δεδομένων Safe Harbor Λόγω της αυξανόμενης σημασίας της ροής δεδομένων, έχει σημασία η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, την ε, πληροφορική της, την διαδικτυακή της ανεξαρτησία και την ασφάλεια της στον κυβερνοχώρο να την καταστήσει μια πρώτη προτεραιότητα και εν ώψη της σύναψης συμφωνιών με τρίτες χώρες όπως η της. Θυμίζω ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα έχει την εξουσία ή όχι να εγκρίνει την τελική συμφωνία διότι όπως και για τη συμφωνία TTIP Είμαστε ένα σώμα δημοκρατικά εκλεγμένο και ε, θα έπρεπε να έχουμε την τελευταία λέξη. Πρέπει λοιπόν να καθησυχάζονται κατά αυτόν τον τρόπο οι πολίτες. Επίσης, οι κανόνες ε, για το δίκαιο, το δικαίωμα μάλλον προστασία των προσωπικών δεδομένων του ιδιωτικού βίου και τη προστασία ε, τη εξορρόπησης επαγγελματικού βίου και ιδιωτικού ε, καταρτίζονται στην χάρτα και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλε τι συμφωνίες με τρίτες χώρε. Επίσης να επιμένουμε στο γεγονό ότι επειδή θα υπάρχει και κυκλοφορία φυσικών προσώπων για την παροχή υπηρεσιών εξαιτία τη συμφωνία τη, θα πρέπει να είναι ίση μεταχείριση όλων των Ευρωπαίων πολιτών, ε, είτε βρίσκονται στη δική μα επικράτεια, είτε στην επικράτεια των υπόλοιπων συμβαλλωμένων μερών. Θα φροντίσουμε να υποβάλουμε τι ανάλογε τροπολογίε για να ληφθούν υπόψη αυτέ τι παρατηρήσει. Πρόεδρο, ευχαριστούμε κύριε Μισελ. Η κυρία Σπινέλη. Μπάρμπαρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τη γνωμοδότηση του συναδέλφου Άλμπρεχτ τη βρίσκω άριστη. Απλώς να τον ρωτήσω πώς προτίθεται να καλύψει αυτήν την τελευταία εξέλιξη, την απόφαση Φρέμς, στην έκθεση του. Διότι η απόφαση ακόμα δεν είναι παραπρόσφατη σε ό,τι αφορά τις αναδυόμενες χώρες κάτι που περιπλέκει κάπως τις διορματεύσεις ήθελα να ρωτήσω πώς θα καλύψει κάποια σημεία ζωτική σημασία για κάποιες χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα όπως η Ρίτρα Ράτσετ. που επιτρέπεται η συνέχιση του δικτυσιακού καθεστώτο των επιχειρήσεων. Δηλαδή, από τη στιγμή που ιδιωτικοποιείται μια εταιρεία, δεν μπορεί να υπάρξει αναστροφή. Αυτό, λόγω των δεδομένων συνθήκων της σημερινής κρίσης, δεν μου φαίνεται σωστό. Θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα αναστρεψιμότητα μια τέτοια απόφαση να μην παραμένει κανείς ε, δέσμιος αυτής της ε, ρήτρας Ράτσετ. Ε, κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η δική μας σκιώδης δεν είναι εδώ σήμερα το απόγευμα, οπότε εκ μέρους της να επισημάνω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, να πω κάτι από προσωπική μου πλευρά. Με όλε τι ε, συζητήσει που έχουμε για τι συμφωνίε ΣΥΤΑ και ΤΙΤΙ, να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι λιγότερο σημαντική ούτε η συμφωνία τη. Αν μην πω ότι είναι ακόμα πιο σημαντική, δεδομένων των συνεπειών που αναμένατε να έχει. Οπότε θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί για το τι κάνουμε εδώ. Σε γενικέ γραμμέ, από τη δική μα την ομάδα, στηρίζουμε πλήρω το σχέδιο ομοδότησης του εισηγητή. Όλο ιδιαιτέρω Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να αντιταχθούμε στις αρχές για την προστασία προσωπικών δεδομένων στο σχέδιο κεφαλαίου που έχουν υποβάλει οι ΗΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο για τι διαπραγματεύσεις. Υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων και με τη συζήτηση που μόλις είχαμε εδώ στην Επιτροπή μας, αλλά και λόγω του χάρτη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι πολύ σημαντικό η προστασία των ιδιωτικών, του ιδιωτικού βίου, η προστασία των προσωπικών δεδομένων να θεωρηθούν εξαιρετικά σημαντικοί τομεί. Υπάρχει ένα είδο προστατευτισμού στην ε, προστασία των προσωπικών δεδομένων και βεβαίω θεωρούμε και θα ε, συνεχίσουμε να διεκδικούμε το απόλυτο δικαίωμα να μοθετούμε σε αυτόν τον τομέα, σε αυτό το πεδίο, όποτε θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο. Θα το επαναλάβω λοιπόν. Συμφωνούμε απολύτω με τον εισηγητή σε όσα προτίθεται να κάνει για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Και τώρα η Επιτροπή. Όχι, Άννα. Συνάδελφοι, παρακαλώ σύντομα στα σχολεία σας. Πολύ σύντομα θα συμφωνήσω απολύτω με όσα είπαν οι προηγούμενοι ομιλητέ, ιδίω ο εισηγητής μα, αλλά να τονίσω ότι και κάτι ακόμη θα πρέπει να τονιστεί, να υπογραμμιστεί εδώ στην όλη συζήτηση και στο σχέδιο νομοδότηση προ την Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου που είναι καθήλυνα αρμόδια. Το ASDS, ο μηχανισμό επιλυση Διαφορών Επενδυτού κράτου. προβλέπει ένα τέτοιο μηχανισμό ε, όπω και η TTIP και η Συμφωνία TISA. Θα πρέπει να το δούμε και να το διαγράψουμε. Πρόεδρο. ο κ. Μπόρνη εκ μέρου τη κυρία Χολμάγερ που ήταν ε, η συγκήτρια του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Αντικαθιστώ την κυρία Χολμάγερ σήμερα. Πολύ σύντομα λοιπόν να σας ενημερώσω ότι το ΕΛΚ εγκρίνει τη συμφωνία τη. Συμφωνεί με το σχέδιο γνωμοδότησης του εισηγητή. Ευχαριστούμε Γιάννη για την έκθεση και απλώς θα θέλαμε μια ελαφρά τροποποίηση στο τμήμα που αφορά την πρόσβαση τα έγγραφα. Θα πρέπει, πιστεύουμε, ε, να παραμείνουμε στην αρχική διατύπωση και να μην αποδεχτούμε τροπολογίες που ε, βγαίνουν εκτός πεδίου της νομοδότησης ή προσπαθούν να χειραγωγήσουν ε, το περιεχόμενο της χρηματοδότησης για άλλους πολιτικούς σκοπούς. Γιατί καταλαβαίνω τώρα από την πίεση των γεγονότων και με την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τον ασφαλή Σίγουρα πρέπει να μελετήσουμε την ε, περίπτωση αυτή, το ασφαλώς λιμένα μεν, αλλά δεν είναι τόσο καλό για την γνωμοδότηση αυτή να προσθέσουμε όλα όσα μπορούν να περάσουν από το μυαλό μας σε αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Μπόνη, η Επιτροπή τώρα. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Η διαπραγματεύσει τη ε, λαμβάνουν ε, χώρα αυτή την εβδομάδα κιόλα. Οπότε να με συγχωρείτε από διευθυντή μου δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα. Όμω εκείνο και οι υπόλοιποι συνεργάτε μα είναι αυτή τη στιγμή στη Γενέβη για να ε, θα φροντίσω να του μεταφερθούν τα ζητήματα που ανέφεραν οι βουλευτέ, έστω και διμερό. Τώρα, οι υπηρεσίε είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα τη οικονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. 70% του ΑΕΠ είναι αυτό που εκπροσωπούν και ε, επίση και ο τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει μεγάλο ρόλο να διαδραματίσει εδώ, με πολύ μεγάλη εξαγωγημότητα ε, και ε, για το εμπορικό μας ισοζύγιο μεγάλη σημασία. Είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί στι υπηρεσίε και θα, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε περισσότερε θέσει εργασία αν ανοίγαμε και άλλε αγορέ για τι υπηρεσίε μα. Διότι οι ευρωπαϊκέ εταιρείε υπηρεσιών έχουν να αντιμετωπίσουν πολλού σημαντικού ε, εμπορικού φραγμού στο εξωτερικό. Γι' αυτό Εάν μπορούσαμε να καθορίσουμε ισότητα στους κανόνες ανταγωνισμού για όλους τους φορείς, αυτό ήταν πολύ καλό για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας στην απασχόληση σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό παίρνουμε μέρος στις συνομιλίες για τις εμπορικές συναλλαγές σε υπηρεσιών. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την Ένωση, θέλουμε να υπάρχει αυτή η πολυμερής συμφωνία και εάν γίνεται στο κατάλληλο πλαίσιο, σε αυτό που τη αρμόζει του ΠΟΕ. Για το σχέδιο γνωμοδότησή σα, ευχαριστούμε για τι παρατηρήσει για τη ροή δεδομένων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα είδαμε και με το ψήφισμα για, το, για τη συμφωνία TTIP. Σίγουρα ε, σωστά, κάποια μέλη έχουν σωστά υποβάλει τροπολογία για τη διασυνορία κυρίων πληροφοριών και να, για να υπάρχουν κάποιε συγκεκριμένε προποθέσει, αλλά σε γενικέ γραμμέ πρέπει να πω ότι στόχο των συστημάτων είναι να μην επιτρέπονται τα διακριτικά και προστατευτικά μέτρα που είδαμε να αναπτύσσονται σε χώρε όπω η Κίνα, η Ρωσία. Και ενώ δεν υπάρχει για την ώρα συμφωνία, ελπίζουμε ότι η Κίνα κάποια στιγμή θα αλλάξει αυτές τις, ε, αυτούς τους κανόνες. Η συμφωνία της βέβαια μπορεί να προβλέπει και μια σειρά από εξαιρέσεις, όπως για την προστασία και το απόλυτο των δεδομένων. Όμως ο βασικός σκοπός των γενικών εξαιρέσεων είναι να επιτρέφουν κάποια μέρη που συμβάλλονται σε μια συμφωνία να ε, επιδιώξουν θεμητούς εμπορικούς σκοπούς ε, με τρόπο λογικό και καλή πίστη. Άρα, σκοπός των εξαιρέσεων δεν είναι να ε, διευρύνουν εξέλεγκτα το πεδίο. Το είδαμε με μερικά μέτρα που επιτράπηκαν λόγω των ε, συμφερόντων ε, της προστασίας της εθνικής ασφάλειας και τάξης λόγω χάρη και επιτρέπουν να διαφύγει κανείς των γενικών του υποχρεώσεων και καθηκόντων. όπως και στην περίπτωση TTIP, λοιπόν, να σας διαβεβαιώσω ότι σε ό,τι αφορά τα πρότυπα προστασία των προσωπικών δεδομένων, αυτά δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων ούτε με αφορμή την συμφωνία ΤΙΖΑ ούτε με καμία άλλη εμπορική συμφωνία. Η συμφωνία ΤΙΖΑ λοιπόν δεν θα αποτελέσει εξαίρεση, δεν θα δημιουργήσει προηγούμενο για να ε, ε, ταράξει το καθεστώς που ισχύει για την προστασία των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο στοιχείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη σχετική ρήτρα. Βεβαίως τις ε, αρχές αυτές τις έχουμε ως προτεραιότητα σε οποιαδήποτε πολιτική ή εμπορική συμφωνία Όμως έχει μια ιδιαιτερότητα η συμφωνία της Είναι μια πολυμερής συμφωνία και τέτοιες ρήτρε όπως τη συμφωνία για τους δημόσιους διαγωνισμούς, τη συμφωνία για τις τεχνολογικές πληροφορίες και τα περιβαλλοντικά προϊόντα, τέτοιες ρήτρε τις προβλέπουμε. Εάν θέλουμε λοιπόν να επανέλθει στους κόλπους του ΠΟΕ στο μέλλον η συμφωνία ΤΙΖΑ, θα πρέπει μια τέτοια ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα να τη σκεφτούμε πολύ σοβαρά, γιατί μπορεί αυτό να αποτρέψει άλλους που σκέφτονται να συμβληθούν ε, να έρθουν προς την κατεύθυνσή μας και βεβαίως να μην πάει καν στο επίπεδο του ΠΟΕ, η Συμφωνία Τίζα. Πάντως, ε, για τις παρατηρήσεις όλων, Βεβαίω θα φροντίσουμε να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση κατά των Ευρωπαίων πολιτών και σας διαβεβαιώνω ότι ούτε στη συμφωνία ΤΙΖΑ γίνεται κουβέντα για έναν μηχανισμό ISDS ως μέρος αυτής. Ολοκληρώνοντας να πω ότι βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις από όσο χρειαστούν και αυτή την εβδομάδα και στην συνέχεια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ τους ε, συναδέλφους και, τον, ε, και τους Κιώδης και Άλμπρε, κύριε Άλμπρε, αν θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Κλωτ. Συνήθως δεν χρειάζεται να επανέλθω, αλλά τέθηκαν κάποια ερωτήματα και θα ήθελα να απαντήσω. Καταρχάς, όσον αφορά την απόφαση του ασφαλούς λιμένα και τον αντίκτυπο τη σε αυτήν την γνωμοδότηση. Δεν πρόκειται απλά για επιθυμία, είναι απέτηση του Κοινοβουλίου στη συμφωνία TTIP και στη συμφωνία Τίσα. να υπάρχει οριζόντια ρήτρα που να βασίζεται στη, στο άρθρο 14 της ε, συμφωνίας ΓΑΤΣ ε, σχετικά με το ε, ανέγκυχτο της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα. δεδομένα μπορούν να τύχουν, ε, θα πρέπει να αφορούν ε, οι συμφωνίες αυτές σε την προστασία των δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και την, κατά τη διαβίβαση σε τρίτες χώρες. Οι δικαστές στο Λουξεμβούργο ξεκαθάρισαν ότι δεν είναι θέμα δικής μας διακριτικής ευχέρειας να παρεμερίσουμε το θέμα αυτό. Αποτελεί απέτηση του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και αποτελεί μέρος της νομοθεσίας μας που βασίζεται στον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν μπορεί λοιπόν να αποτελεί μέρος των διαπραγματεύσεων μια επιδείνωση των κανόνων. Επιτρέψτε μου επίσης να προσθέσω ότι όσον αφορά τον τόπο των δεδομένων ε, είναι και αυτό σχετικό θέμα. Αν χρειάζεται να γίνει επεξεργασία των δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε δεν επιτρέπεται μια εμπορική συμφωνία να υπονομεύσει αυτόν τον κανόνα, ούτε επιτρέπεται να αναγκάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαβιβάσει αλλού δεδομένα ε, παρά τη, σε αντίθεση με την ομοθεσία της. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά προδικάσαμε αυτό που είπε ε, και το δικαστήριο όσον αφορά το ISDS στην ανακόμεση να πω ότι στην ΤΙΣΑ δεν προβλέπεται ε, τέτοιος μηχανισμός, δεν χρειάζεται λοιπόν ε, να αγωνιστούμε για αυτό το θέμα. Όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα, σημειώνω την επιθυμία του ΕΛΚ. Πολύ θα ήθελα και συγκεκριμένη πρόταση, αν πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει το κείμενο, εάν θέλουμε να συμφωνήσουμε ε, πάνω στην γνωμοδότηση ε, όπως ψηφίστηκε. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν ενωμένοι. Τέλος, σε μια σύντομη παρατήρηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προσεκή παρατήρηση. Δεν νομίζω ότι βρίσκεται στη διακριτική ευχαίρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεπουλήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ίσως δεν κατάλαβα καλά αυτά που είπατε σχετικά με την προσχώρηση άλλων χωρών στην ΤΙΣΑ ε, εφόσον υπάρχει ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, θα ήθελα να σας προειδοποιήσω ότι μπορεί έτσι να οδηγηθούμε σε ε, ασυνετή στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις ρήτρες αυτές στις διεθνείς συμφωνίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. 16 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 19η Οκτωβρίου. Το επόμενο μας θέμα είναι η κατάσταση των ε, τριμερών διαπραγματεύσεων για την προστασία των ε, φυσικών ε, προσώπων εναντί της επαξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Έχεις λοιπόν το λόγο πάλι Ευχαριστώ πολύ θα σας ενημερώσω σχετικά με την πρόοδο των τριμερών διαπραγματεύσεων. Είναι δεύτερη φορά που σας ενημερώνω σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον Ιούλιο. Μετά την συμφωνία του Συμβουλίου πάνω στην γενική προσέγγιση για τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων. Όπως είπα νωρίτερα, καταφέραμε πριν το καλοκαίρι, οι διαπραγματεύσεις για το κεφάλαιο 5 να ολοκληρωθούν που αφορούν ε, την ε, διαβίβαση σε τρίτες χώρες. Και είχαμε πει ότι αν το δικαστήριο εκδώσει απόφαση για τον ασφαλή λιμένα πριν την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, μάλλον θα πρέπει να επαναξετάσουμε κάποια θέματα. Οπότε μάλλον έχουμε φτάσει στη στιγμή που η διαπραγματευτική ομάδα θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά την απόφαση και να δει σε τι βαθμό είναι απαραίτητο να επαναδιαπραγματευτεί κάποια συγκεκριμένα θέματα στο κεφάλαιο 5. Γενικά πάντως νομίζω ότι έχουμε σημειώσει πρόοδο μετά τις θερινές διακοπές. Επανήλθαμε, συνεχίζουμε να καταβάλουμε σημαντικές προσπάθειες, ε, καθότι είναι τεράστιο νομοθετικό πακέτο. Ασχολούμαστε με τα δικαιώματα των ατόμων αλλά και τις υποχρεώσεις ε, και τα καθήκοντα των ε, ελεγκτών. Τα κεφάλαια 2, 3 και 4 έχουν εξεταστεί στις τριμερείς διαπραγματεύσεις και μετά από τις συναντήσεις που είχαμε υπολογίζω ότι έχουμε πετύχει συμφωνία στο 70 με 80% αλλά δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Υπάρχουν κάποια θέματα, κάπως πιο πολιτικά, όπου υπάρχουν διαφορές ε, ανάμεσα στις ε, διάφορες διαπραγματευτικές εντολές. Θα πρέπει να επανέλθουμε στα θέματα αυτά. Να σας αναφέρω κάποια από τα θέματα. Για παράδειγμα, η μορφή και οι προϋποθέσεις της ε, συγκατάθεση ατόμων για την επεξεργασία δεδομένων. Το κατά πόσο η ελαχιστοποίηση των δεδομένων ε, θα ορίζεται και θα ρυθμίζεται στο κείμενο και επίσης η συγκεκριμένη διατύπωση των υποχρεώσεων για την σωστή ενημέρωση ατόμων σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Ε, διαπραγματευόμαστε λοιπόν ε, ακόμα το θέμα αυτό καθώς και τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των ελεγκτών. Θέλουμε λοιπόν να εναρμονίσουμε το ζήτημα του διορισμού υπεύθυνου για την προστασία των δεδομένων, όπως ζητάει το Συμβούλιο από τα κράτη-μέλη. Εδώ είχαμε κυρίως διαφορά στις διάφορες προσεγγίσεις, αλλά μπορώ να σας πω ότι σε πολλά ζητήματα, βρισκόμαστε πολύ κοντά στις θέσεις μας ή ακόμα και συμφωνούμε. Θα λύσουμε λοιπόν τα απλά θέματα για να φτάσουμε στα πιο πολύπλοκα. Η ευελιξία μας ε, όσον αφορά την προσέγγιση των θέσεών μα σε αυτές του Συμβουλίου εξαρτάται από τους σκιώδεις συζητητές. Είναι σημαντικό να θυμίσω σε όλες τις πολιτικές ομάδες ότι θα πρέπει να ενημερώσουν τα μέλη τους ώστε η διαπραγματευτική ομάδα να μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται με βάση την εντολή που έχει δοθεί σε αυτήν και τις απόψεις των πολιτικών ομάδων. Νομίζω ότι είναι δυνατόν να ολοκληρώσουμε μια συμφωνία με το Συμβούλιο μέχρι το τέλος της χρονιάς, όπως προβλέψαμε, και τα τρία θεσμικά όργανα κατά το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων. Θα επανεξετάσουμε τις εκκρεμότητες κατά διάρκεια του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου. Θα συνεχίσουμε την πρόοδό μας, ε, διότι ε, στις διαπραγματεύσεις θα φτάσουμε τώρα στα κεφάλαια 6 και 7. Θα εξετάσουμε δηλαδή τη συνεργασία μεταξύ των αρχών προστασίας των δεδομένων στα 28 κράτη-μέλη. Θέλουμε ε, ενιαία και ε, συνεκτική εφαρμογή των κανόνων. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη ε, και πιο συνεπή επιβολή του νόμου. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε σύντομα τα θέματα αυτά, διότι προσεγγίζουμε ο ένας τις θέσεις του άλλου, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, και θα φτάσουμε στο θέμα των κυρώσεων. Αλλά και πιο σημαντικό είναι ότι θα αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για την οδηγία για την προστασία των δεδομένων και έτσι θα ξεκαθαριστεί και το πεδίο εφαρμογή των δύο νομοθετικών μέσων που θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης όταν ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις και για την οδηγία για την προστασία των δεδομένων. Αυτά από μένα. Είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ, Γιάν. Αναρωτιέμαι αν οι σκιώδεις συζητητές θα θέλουν να πάρουν το λόγο. Παρακαλώ η κυρία Λόριστην. Θα ήθελα πολύ σύντομα ε, να σας ενημερώσω σε συνέχεια αυτόν που, που είπε ο Γιάννο ότι βρισκόμαστε στην αρχή των διαπραγματεύσεων για την οδηγία. Σήμερα είχαμε την πρώτη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών και διατηρούμε την προσέγγιση που είχαμε στο πακέτο αυτό και ακολουθούμε την ίδια οδό και στο, στον κανονισμό και στην οδηγία. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις προς τον Γιάννα Άλπρεχτ. Όχι. Σημειώνω αυτό που είπε ο Γιάννος όσον αφορά την ε, ανοιχτή του θέση απέναντι στις ε, πολιτικές ομάδες. Ε, θα πρέπει να ληφθούν πολλές πολιτικές αποφάσεις. Είναι πολύ έντονος ο τριμερής διάλογος. Γνωρίζω πολύ καλά την ε, δουλειά που γίνεται, διότι πραγματοποιούνται και ταυτόχρονα πολύ τριμερείς διάλογοι. Θα ήθελα λοιπόν να τον επενέσω για αυτό που είπε. Θα είναι σημαντικό λοιπόν να προσέξουμε τα σημαντικά θέματα που θα πρέπει να τοπίσουμε κατά τη διάρκεια των τριμερών διαλόγων. Αλλά όλοι αυτοί οι τριμερείς διάλογοι δείχνουν πόση δουλειά έχει η Επιτροπή μας. Σε ευχαριστώ Ιάν. Και έχουμε άλλη μία έκθεση για την ε, οποία έχουμε τριμερείς διαπραγματεύσεις. Ε, ίσως να αναβάλουμε λίγο το θέμα διότι έρχεται, ε, καταφάνει ο εισηγητής, ο κύριος Κερτχόπ, όταν έρθει θα μπορέσουμε να συζητήσουμε το θέμα των ε, δεδομένου έρχονται στου φακέλους επιβατών. Αν δεν έχετε αντίρρηση θα προχωρήσουμε στο σημείο 8, λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές Δημόσιε διοικησει τι επιχειρήσεις και τους πολίτες. Κύριε Λενάρς, θα μας παρουσιάσετε την πρόοδο των, τριμερών διαπραγματεύσεων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Επτά τεχνικές ε, συνεδριάσεις είχαμε στον τριμερή διάλογο και έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει ε, τη συζήτηση. Ήταν πολύ σκληρέ οι διαπραγματεύσεις, πρέπει να σας πω, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, τα θέματα που άπτονται της δικής μας Επιτροπής. Από πλευρά Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είχαν ξετρελαθεί, για να το πω έτσι, να συνεργαστούν και να συμπεριλάμουν τις δικές μας τροπολογίες που ε, είχαμε εισαγάγει εμείς στην έκθεσή μας. Πάντως τελικά ήταν πολύ καλό το αποτέλεσμα πρέπει να πω. Χάρη μεταξύ άλλων και στις προσπάθειες των συναδελφών της Επιτροπής ε, Ήτρε που είχαν και την ευθύνη των διαπραγματεύσεων ε, και υποστήριξαν τις δικές μας θέσεις. Έχουμε μία αιτιολογική σκέψη για την προστασία των δεδομένων στο κείμενο, πολύ εκτενές και ένα άρθρο νέο για την προστασία των δεδομένων στο κείμενο των άρθρων και όχι σε αιτιολογικές σκέψεις. Και η προστασία των δεδομένων και η ιδιωτική ζωή είναι σημαντικές ε, ε, ξεχωριστές ειδικέ αρχές του κειμένου. Αυτά είναι τα βασικά. Στην αιτιολογική σκέψη επίσης αναφέρουμε ε, στις ε, λύσεις διαλειτουργικότητας και την εξασφάλιση της προστασίας ε, των δεδομένων θα πρέπει να είναι κάτι το ε, γενικό και ο κανόνας. Και η προστασία των δεδομένων βεβαίως εντάσσεται και στον κανονισμό και από εκεί και πέρα ό,τι εκπονείται ή ε, εντάσσεται στο πρόγραμμα ίσα για τη διαλειτουργικότητα λαμβάνει αυτά τα θέματα υπόψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους συνεισέφεραν στην προσπάθειά μας. Ευχαριστώ. Ξέρω ότι προσπαθείτε να προβάλλετε πάντα και να φέρετε στο προσκήνιο τα θέματα της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν έχουν ερωτήσει άλλοι συνάδελφοι για τη διαλειτουργικότητα. Όχι. No, that... so Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση αυτή. Δεν ξέρω ήρθε ο κύριο Κίρκοπ. Ή να πάμε στο σημείο 9. τον εισηγητή μας για ε, τους φακέλους επιβατών, το PNR. Στο μεταξύ μπορούμε να ασχοληθούμε με τον ΕΝΕΑ. Fortunately, Ευτυχώς είναι εδώ ο κύριος Γέτζεκ. So this is the... Ε, ετήσια έκθεση 2014 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερών της Ένωσης, κατά πολέμηση της απάτης. Ο Πίτερ Γέζεκ ε, των Φιλελευθέρων είναι ε, συντάξει της γνωμοδότησης. Αν θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τον ελέγχουν φαίνεται τον κύριο Κίρκοπ στα εσωτερικά σύνορα της Ένωσης, γι' αυτό καθυστερεί. Ας μιλήσω εγώ τώρα λοιπόν μέχρι να έρθει για την καταπολέμηση της απάτης. Αυτό που με ενδιαφέρει κυρίως είναι τα εξής δύο. Πρώτον, Πρόσφατα ελήφθησαν πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να προστατευτούν τα συμφέροντα, τα οικονομικά της Ένωσης. Όπως γνωρίζετε, το 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε δύο ε, μέσα για το ποινικό δίκαιο και τα δύο στοχεύουν στην ενίσχυση της ε, προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, πάντα για το ποινικό δίκαιο αναφέρομαι. Το, η πρώτη είναι η οδηγία, ε, μάλλον η δεύτερη είναι για τον εισαγγελέα και η πρώτη είναι μια αντίστοιχη. Ε, έχει έρθει η ώρα τώρα μαζί με το Συμβούλιο να δώσουμε νέα όθηση ε, για την ε, οδηγία ΠΙΦ. Ε, στο τελευταίο τριμερή διάλογο ε, σχεδόν συμφωνήσαμε για όλα τα θέματα, αλλά τελικά υπήρξε μπλοκή για ένα ζήτημα πολύ κρίσιμο, αν ε, θα συμπεριληφθεί η απάτη για το ΦΠΑ. Το διαφυγόν και εδώ ε, για την Ένωση είναι 168 δισεκατομμύρια ευρώ παρακαλώ από την απάτη στο ΦΠΑ. Είναι πολύ σημαντικό για τα κράτη-μέλη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμφωνήσουν για τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορεί να, λυθεί αυτό το μείζον πρόβλημα. Ε, δεύτερον, το σχέδιο γνωμοδότησής μου βασίζεται στην ανάγκη συνέχισης ε, για την καταπολέμηση της διαφθοράς που εκτιμάται ότι κοστίζει στα κράτη-μέλη 120 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως παρακαλώ πέρσι το Φεβρουάριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, ε την πρώτη της έκθεση κατά της διαφθοράς και ήταν για μένα πολύ καλό πρώτο βήμα μόνο. Ε, είχαμε πλήρη ε, εικόνα σε όλα τα κράτη-μέλη ε, για την κατάσταση και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Η έκθεση αυτή έδειξε ότι παρόλο ε, που διαφέρει από κράτος σε κράτος το επίπεδο της διαφθοράς, αφορά όλα τα κράτη-μέλη Και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους θεωρούν ότι η διαφθορά στη χώρα τους αυξήθηκε την περασμένη τρία ετία. θέλουμε αν θέλουμε μάλλον να είμαστε αξιόπιστοι στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης, θα πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα σε ό,τι αφορά την ακαιρεότητα, τη διαφάνεια για τις συγκρούσεις συμφερόντων, όπως αναμένουμε άλλωστε και από τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό στην γνωμοδότησή μου καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει ειδικό κεφάλαιο για τις επιδόσεις των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στην καταπολέμηση της διαφθοράς στη δεύτερη έκθεση κατά της διαφθοράς που αναμένεται να εκδοθεί στην αρχή του 2016 και όχι αργότερα. Για να ολοκληρώσω, αυτά είναι τα δύο βασικά καινούρια δικά μου σχόλια για τη γνωμοδότηση και θα ήθελα χαρά να ακούσω και τους σκιώδεις ε, ε, συγγητές. Ευχαριστώ. Δεν είμαι βέβαιο. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μεταφέρω το μήνυμα του συναδέλφου Μακοβέη που λέει ότι για τον εισηγητή από το, για τον κύριο Γέζεκ πρέπει να πω για τις ευρωπαϊκές οδηγίες ότι θα πρέπει να δράσει με αποφασιστικότητα το Κοινοβούλιο και όχι μόνο να δώσει νέα όφεση στην εξέταση του θέματος αυτό αλλά να παρατρύνει το Συμβούλιο να οδηγήσει σε ολοκλήρωση τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει να είναι αυτό ένα σημαντικό πεδίο όπως ε, επισημαίνει ο εισηγητής το θέμα του ΦΠΑ που οδηγεί σε απολύες 2 δις ευρώ ετησίω λόγω τη μη καταλληλότητα του συστήματο. Θα πρέπει λοιπόν να περιλαμβάνεται υπόψη σε όλε τι συναλλαγέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω τη τωρινή κατάσταση, αν τα χρήματα των φορολογουμένων θεωρούνται ισότιμα παντού και αν ένα κατοσμέλο δεν κάνει τη σωστή ε, ε, διερεύνηση ή κατάσχεση, χάνουν όλοι μα οι πολίτε. Επίσης, τονίζουμε προς τον εισηγητή ότι θα πρέπει να δώσουν το παράδειγμα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και να ακολουθούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα για τη διαφάνεια, την ε, ε, συγκέντρωση δεδομένων και τις συγκρούση συμφερόντων. Όμως, προκειμένου να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρχουν διεξοδικά κριτήρια για την καταπολέμηση της διαφθοράς και να ισχύουν και για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ιδίω στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων. Αυτέ είναι οι παρατηρήσει τη κυρία Μακοβέη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Um, Ευχαριστώ, κύριε που μας μεταφέρατε την τοποθέτηση της κυρίας Μακοβέη για σας είπε ο κύριος Γέζεκ. Κύριε Γέζεκ, έχετε να πείτε άλλα πράγματα. Αλλιώς μπορούμε να κλείσουμε. Πολύ σύντομη αντίδραση, Πρόεδρε. Εάν βρούμε τρόπο να παρατρύνουμε το Συμβούλιο να αναλάβει δράση με τα χαράς, αλλά νομίζω ότι στην όλη διαδικασία που με του κοιόδε θα τα καταφέρουμε. Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Οι προθεσμοί του για τι τροπολογίε είναι στι 14 Οκτωβρίου και 1 Δεκεμβρίου στι 11 Νοεμβρίου και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μα 1 Δεκεμβρίου. Και τώρα για το Ευρωπαϊκό Αρχείο Επιβατών. Τη γιατί είναι ο κ. Κίρκοπ. και θα μας παρουσιάσει το τι έγινε στον πρώτο γύρο του τριμερούς διαλόγου 24 Σεπτεμβρίου και 29 Σεπτεμβρίου στο δεύτερο γύρο. Κύριε Κίρκοπ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως όλοι γνωρίζετε. Θα υιοθετήσουμε, υιοθετήσαμε την ε, θέση της ΛΥΜΠΕ για το θέμα αυτό πριν ε, το καλοκαίρι. Ξεκινήσαμε, όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, τον τριμερή διάλογο τον Σεπτέμβριο και ε, συνεχίζονται οι συζητήσεις. Θα ήθελα να ξανατονίσω ότι το Κοινοβούλιο μας έχει δεσμευτεί να ολοκληρώσει το θέμα αυτό μέχρι το τέλος της χρονιάς και αυτό συνεχίζει να είναι ο στόχος μου. Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμερούς διαλόγου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε την ανάγκη να υιοθετηθεί έγκαιρα η οδηγία αυτή και 14 κράτη-μέλη έχουν αρχίσει να ετοιμάζουν τεχνικά εθνικά τους συστήματα αυτή τη στιγμή. Μετά από 3,5 χρόνια ε, δεν θα μπορούσα να υποστηρίξω ότι η ταχύτητα είναι το μόνο μας κριτήριο εδώ. Αλλά Πολλά κράτη-μέλη δεν έχουν τα απαραίτητα συστήματα για να χειριστούν τα δεδομένα που περιέχονται στους ε, φακέλους επιβατών. Κατά τον πρώτο τριμερή διάλογο διαπιστώθηκε ότι τα τρία θεσμικά όργανα είχαν διστάμενες ε, απόψεις και ε, το ε, διεθνές ε, έγκλημα ήταν το βασικό πρόβλημα και οι συζητήσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες και είμαι αισιόδοξο ότι το πνεύμα του συμβιβασμού θα επικρατήσει. Άλλες συζητήσεις είχαν να κάνουν με τους οικονομικούς φορείς που θα καλύπτονται από την οδηγία αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πραγματοποιήσει διάσκεψη για ε, τα δεδομένα PNR, όπου θα συζητηθεί και το θέμα αυτό. Επίσης, ε, θέμα ήταν ε, οι πτήσεις. Δεν θεώρησα ότι ήταν απαραίτητο να γίνει σχετική συζήτηση με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχω δώσει τον λόγο στους Ευρωβουλευτές ότι θα έφυγα το θέμα. Στις 29 Σεπτεμβρίου συζητήθηκαν τα άρθρα 6 και 11. Στα άρθρα αυτά τα θεσμικά όργανα ε, κατάφεραν να συμφωνήσουν σε περισσότερα θέματα. Όσον αφορά όμως ε, τις μονάδες ε, πληροφόρησης των επιβατών που ενημερώνουν τους επιβάτες σχετικά με τα δικαιώματά τους και πώς μπορούν να τα ασκήσουν, ε, συζητήθηκε αν είναι απαραίτητες αυτές οι μονάδες ή ε, αν ε, αποτελούν ένα περιττό γραφειοκρατικό άκτος καθότι δεν έχουν άμεση πρόσβαση στους επιβάτες. Επίσης συζητήθηκε το θέμα της λογοδοσίας των μονάδων ενημέρωσης των επιβατών. Θα συνεχιστούν οι συζητήσεις. Κατόπιν είχαμε τα ε, άρθρα 4 και 11 που έχουν να κάνουν με την εμπιστευτικότητα των ε, δεδομένων. Ε, σημαντικό θέμα εδώ ήταν η διάκριση ανάμεσα στις εμπορικές δραστηριότητες των εταιριών αερομεταφορών και τις διατάξεις της οδηγίας PNR και έχουμε και θα πρέπει να φροντίσουμε να μην προκαλεί σύγχυση η σχέση ανάμεσα στην οδηγία PNR και την οδηγία 9546 και να μην ε, τιμωρούνται διπλά οι ε, ε, αεροπορικές εταιρείες. Όσον αφορά το διάστημα διατήρησης των δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 9, το Συμβούλιο έχει διαφορετική άποψη. Το κλήθηκε το Συμβούλιο να παρουσιάσει στοιχεία στο Κοινοβούλιο και την Κομισιόν ε, σχετικά με το γιατί θα πρέπει να απομακρυνθούμε από τις ε, διατάξεις που προτείνει η Κομισιόν και τη θέση που έχει υιοθετήσει το Κοινοβούλιο. Ε, στόχος του Κοινοβουλίου ήταν να αποφύγουμε περαιτέρω κατακαιρματισμό. Ωστόσο, το Συμβούλιο έχει διαφορετική θέση και είναι υπέρ μιας λιγότερο αυστηρής προσέγγισης. Ε, μία από τις ανησυχίες του Συμβουλίου έχει να κάνει με τις διαφορές ε, με την ε, νέα οδηγία προστασίας δεδομένων. Ωστόσο το Κοινοβούλιο όμως έχει καταστήσει σαφές ότι θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων των επιβατών για να προστατευτούν σωστά τα δεδομένα αυτά. Επίσης, ε, το Συμβούλιο υποστηρίζει ότι αν δεν συμπεριλαμβάνονταν οι εσωτερικές πτήσεις, αυτό ε, θα ήταν η βάρος της ασφάλεια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, δεδομένου ότι το 80% των δεδομένων που συλλέγουν κάποιες εταιρείες αφορά εσωτερικές πτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κοινοβούλιο ζήτησε περαιτέρω πληροφορίες πάνω στο θέμα αυτό. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι στο θέμα αυτό το Κοινοβούλιο σαφώς είχε επιλέξει να αποκλείσει τις εσωτερικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θα πρέπει να έχουμε μια εις συζήτηση στο μέλλον πάνω στο θέμα αυτό. Στο μεταξύ έχω ζητήσει από το ε, Συμβούλιο να δώσει στο Κοινοβούλιο και την Κομισιόν ε, περαιτέρω ε, αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαιότητα αυτού. Κύριε Πρόεδρε, βλέπετε ότι έχουμε καλύψει κατά τις δύο πρώτες σε συναντήσεις τριμερούς διαλόγου τα σημαντικότερα θέματα και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε καλό συμβιβασμό. Η επόμενη συνάντηση για τον τριμερή διάλογο θα πραγματοποιηθεί στις 20 Οκτωβρίου ε, και πολύ ευχαριστώ θα ενημερώσω την Επιτροπή ε, αμέσως μετά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε πρώτα τους σκιώδης εισηγητές, η Πίρκη Τσίπελ. Πρόεδρος, ζητώ συγγνώμη κυρία Χολμάιερ, είπατε ότι θέλετε το λόγο. Κακή συνήθεια μου γίνεται. Κυρία Σίπελ, παρακαλώ. Δεν φταίω εγώ, δεν ζήτησα το λόγο. Ε, συγγνώμη, για όσους δεν παρακολουθείτε, μιλάμε για τη σειρά που θα πάρουν το λόγο και όδησες ηγητές. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, ε, θα ήθελα να πω ότι γνωρίζω καλά το θέμα αυτό, διότι συμμετείχα στις διαπραγματεύσεις. Ε, το Κοινοβούλιο ε, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να καταλήξει σε κάποιο αποτέλεσμα εντός του έτους. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι έχοντας κατά νου την απόφαση του δικαστηρίου για τη διατήρηση των δεδομένων και για τον ασφαλή λιμένα, θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την καλή νομοθεσία, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να ευθυγραμμίζεται με τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα μας παρουσιάσει πιο καλά επιχειρήματα, διότι κανένα από τα θεσμικά όργανα δεν θα υποφεληθεί εάν παρουσιάσουμε μια οδηγία την οποία θα ακυρώσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα αναφερθώ σε κάποιες από τις λεπτομέρειες, θα επικεντρωθώ σε κάποια θέματα. Το Συμβούλιο υποστηρίζει και πάλι ότι θα πρέπει να αποφύγουμε ε, το περιττό οικονομικό άχθος για τις εταιρείε αερομεταφορών και για ε, τις μονάδες ενημέρωσης ε, των επιβατών, PIU. Αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί εγώ νομίζω ότι η δημιουργία των PIU με όλες τις τεχνικές απαιτήσεις, ε, με το ε, ειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται, αυτό από μόνο του, νομίζω θα συνεπάγεται υψηλό κόστος. Και κανείς ε, δεν ισχυρίστηκε ποτέ ότι αυτό είναι περιττό άχθος. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να εξετάσουμε την προστασία των δεδομένων υπό το φως της αναλογικότητας και Όσον αφορά τα PIU, υποστηρίχθηκε ότι δεν υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στο PIU και τον επιβάτη. Μα φυσικά υπάρχει άμεση σχέση, διότι επί χρόνια λαμβάνουν τα, προσωπικά μου δεδομένα. Η εταιρεία η αεροπορική εταιρεία δεν μπορεί να ενημερώσει σχετικά με το τι ακριβώς κάνει το PIU με τα δεδομένα μου. Θα πρέπει λοιπόν κάτι να γίνει για το θέμα αυτό όσον αφορά ε, τον ε, επόπτη προστασία δεδομένων. και σε άλλε σχετικέ συζητήσει έχουμε διαπιστώσει ότι ναι, είναι πολύ ωραίο να έχουμε ε, έναν υπεύθυνο προστασία δεδομένων, αλλά θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό φυσικά και θα πρέπει να είναι, διότι εάν είναι προαιρετικό το να δημιουργηθεί αυτή η θέση, μπορώ να σας ε, διαβεβαιώσω ότι ε, κάποια κράτη-μέλη ποτέ δεν θα έχουν επόπτη προστασία δεδομένων και γιατί όχι, εάν όλα γίνουν σωστά, εάν τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας δεδομένων του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, δεν θα υπάρχει λόγος να προσφύγει κανείς και θα μπορεί πάντα από τις προστασίες δεδομένων να μας ενημερώνει ότι όλα πάνε κάνα και όλοι είναι ικανοποιημένοι. Όσον αφορά λοιπόν τις ε, κάποιες ε, πτήσεις ε, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο δικαστήριο θα πρέπει να εξετάσουμε και πάλι προσεκτικά το θέμα αυτό όσον αφορά το ποιες πτήσεις θα καλύπτονται. Ελπίζω λοιπόν ότι όλοι θα έχουμε καταλάβει ότι όλα τα θεσμικά όργανα θα υποφεληθούν αν ε, υιοθετήσουμε όχι έναν οποιονδήποτε νόμο, αλλά έναν σωστό νόμο, καλοδιατυπωμένο και γι' αυτό προσλέπουμε στον επόμενο γύρο του τριμερούς διαλόγου για να σημειώσουμε πρόοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Μόνικα Χολμαϊερ, παρακαλώ. Λοιπόν, πρώτον, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα τον εισηγητή για την εξαιρετική διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων και με εντατικό τρόπο μάλιστα τα φροντίζει αυτά τα θέματα. Προσωπικά θεωρώ ότι και θέλω να ρωτήσω το Συμβούλιο Μπορεί να μας δώσει συγκεκριμένα στοιχεία το Συμβούλιο Πραγματογνωμοσύνη για τις ενδοευρωπαϊκές στήσεις, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς, ποιος, γιατί και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, γιατί για το Σέγγεν Πάντα τονίζεται ότι δεν υπάρχει σχέση, αλλά τονίζεται με αλφαγιώτα. Χρειαζόμαστε όμως ε, και μια νομική γνώμη για το κατά πόσο όλα αυτά συνάδουν με το Σέγγεν και με τις συνθήκες ακόμα. Προσωπικά πιστεύω ότι έχει δίκιο το Συμβούλιο, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει οι νομικές ρυθμίσεις να ε, υποστηρίζονται και με το σωστό τρόπο γιατί μπορεί τελικά να ακυρωθεί μια νομοθεσία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή να υποχρεωθεί κάποιος να την αναθεωρήσει λόγω ανεπαρκούς ε, νομικής βάσης υποστήριξης. Ο εισηγητής πιστεύει ότι θα προλάβουμε να ολοκληρώσουμε το θέμα μέχρι τα τέλη του έτους γιατί άκουσα τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας στο Κοινοβούλιο, τον κύριο Λαντ, που είπε ότι προσοχή, ε, πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με τα θέματα ασφαλείας και να δούμε πώς έχει η σημερινή κατάσταση. Είναι μεγάλες και δύσκολες οι τρομοκρατικές ε, επιθέσεις που γίνονται και υπάρχει μια δυσκολία στο χειρισμό όλης αυτής της κατάστασης. Ε, Γίνεται λόγος για περιττό κόστος ε, για τις ε, υπηρεσίε ενημέρωση των επιβατών, το PIU. Μα κοιτάξτε, εκεί οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι πραγματικά ειδικοί. Αλλιώ τι νόημα έχει. Το βλέπουμε σε διάφορα κράτη-μέλη ήδη ε, που έχουν πιο μακροχρόνια εμπειρία και μου φαίνεται προβληματικό να εξετάζεται αυτό το θέμα αμυγός με όρους κόστους δηλαδή η μείωση προσωπικού, η μείωση εμπειρογνωμόνων ε, δεν θα πρέπει να γίνει για λόγους οικονομίας. Θέλουμε να έχουμε καλό σύστημα πιενά που να λειτουργεί σωστά και να ε, λειτουργεί και στοχευμένα μόνο εναντίον κάποιων ε, σεσημασμένων εγκληματιών. και δεν θα πρέπει να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα επιπόλαια αλλά να δικαιολογούνται και απέναντι στο ε, δικαστήριο. Γιατί υπάρχει ο περιορισμός του προσωπικού να μην είναι μόνο ο λόγος οικονομικός. Χρειάζεται και μια προεργασία υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα τα οποία δεν βλέπει κανείς. Είναι μαθηματικοί αλγόριθμοι και τα λοιπά και καλό ε, είναι να περιορίζονται ακόμα περισσότερο για να εξασφαλίζεται η προταστασία των δεδομένων. Ελπίζω τα κράτη-μέλη να συμφωνούν μαζί μας και να είναι πάρα πολύ ακριβή στην προσέγγιση τους γιατί σε τελική ανάλυση διακυβεύεται και η ε, αποτελεσματικότητα και η προστασία των δεδομένων. Και τα δύο αυτά είναι άψη του ιδίου νομίσματος και για μένα θετικά. Θα ήθελα να μου πει το Συμβούλιο τι ακριβώ γίνεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομη, διότι δεν μπόρεσα να πάρω μέρο στου τριμερεί διαλόγου. Έχουμε περάσει σε μια περίοδο που Πρέπει να είμαστε παρόντε ταυτόχρονα σε τρομερού διαλόγους και συνεδριάσει στι Βρυξέλλε που όλα εκκλείζονται στι Βρυξέλλε ταυτόχρονα. Παρ' όλα αυτά δεν αισθάνομαι ενοχέ. διότι μπορεί να μην συμφωνούμε με τον ε, Τίμωθη σε όλε τι πλευρέ αυτή τη ε, οδηγία, αλλά τον εμπιστεύομαι ότι θα μας εκπροσωπήσει με φιλότιμία και εντυμότητα ως Κοινοβούλιο συνολικά στις δημοκρατήσεις. Ως προς τα αποτελέσματα των, της προφορίας στην ΛΥΜΠΕ δεν νομίζω θα είναι απλό αυτό που έχετε αναλάβει. Ε, θα είναι πολύ περι, στενό το περιθώριο και ίσως το Συμβούλιο να θέλει να συμπεριληφθούν οι εσωτερικές πτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μέρος της εντολής μας. Οπότε σε ό,τι με αφορά δεν υπάρχει καν ανάγκη να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Εάν θέλουν να έχουμε ένα μετρό για τι εσωτερικέ πτήσει να κάνει μια πρόταση. Δεν είναι μέρος τη εντολή. Τόσο απλά. Έπειτα, να είμαστε σαφείς για τη θέση του Συμβουλίου. Και εκεί μιλάμε για θέση πλειοψηφία. κάποιε χώρες δεν συμφωνούν με τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί. Με αυτό λοιπόν το στοιχείο είναι σημαντικό η έκφαση των διπλωματεύσεων, ναι, να είναι αδιάβλητη κατά 100% από νομική άποψη. Να μην υπάρχει καμία δυνατότητα νομική αμφισβήτηση. Γιατί αν μια μη κυβερνητική οργάνωση, κάποιο πολίτη, θέλει να προσφύγει στα τη μέλη, θα μπορεί να το κάνει εάν νομικό δεν είναι 100% ασφαλή η τελική έκβαση. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Να πάμε πάλι πίσω στον ε, εισηγητή. Υπάρχουν αρκετέ ερωτήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έγιναν αρκετέ παρατηρήσει, ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσε, τι σημείωσα προσεκτικά, αλλά δεν πρόκειται να τι απαντήσω τώρα. Ενημέρωσα για το που βρισκόμαστε. Ναι, το βλέπω, αλλά δεν λέμε τώρα εδώ στην απενημέρωση για του τριμμένου διαλόγου που είναι έτσι κι ε, Δεν είναι ένα ένας γύρος απαντήσεων. Απλώ λέω αν θέλετε να πείτε κάτι προ του συναδέλφου, διότι έγινε μια σειρά από ερωτήσει. Ό,τι θέλετε να απαντήσετε. Πρόεδρε, θα έκανα μια γενική παρατήρηση για αυτόν τον λόγο. Για αυτόν τον σκοπό, μάλλον. Ε, καλωσορίζω τι ερωτήσει και είναι μια ευκαιρία να ξαναδούμε πώ έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, αλλά ακόμη η, όλη η συζήτηση είναι υπό εξέλιξη. Υπάρχουν κάποια σημεία λίγο πιο δύσκολα, υπάρχουν κάποια θέματα κάπως πιο ευαίσθητα, τα έφεξε και το ΕΛΚ. Εδώ δεν υποτιμώ τις ευθύνες που έχω στο πώς έχω αναλάβει να χειριστώ το θέμα, αλλά θα είμαι πολύ πρόθυμος και συνεργάσιμος όπως πάντοτε σε τέτοιες διαδικασίες. Υπάρχουν κάποια δύσκολα προβλήματα σε ορισμένα σημεία, το γνωρίζουμε, αλλά σκοπεύω να αποσπάσω κάτι που θα είναι ικανοποιητικό για όλους, θα λειτουργήσει και θα είναι και μια ισχυρή έκβαση, μια καλή έκβαση των διπλωματεύσεων να ολοκληρωθούν. Θα συνεχίσω πάντω να σα ενημερώνω για τον πρόεδρο που αποτελείται. Πρόεδρο, να πω στου συναδέλφου παρόλο που τελειώνουμε να δει και σε όσου παρευρίσκονται ότι είχαμε έξι απενημερώσει για τον διαλόγου σα τώρα. Και όπω είπε και η Σόφη Ιντβελτ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, δείχνει τι μεγάλο έργο έχει αναλάβει η Επιτροπή μα. Θέλω σε κάθε περίπτωση να ευχαριστήσω του συναδέλφου που ε, συμμετέχουν σε αυτέ τι εργασίε υψηλού επίπεδου και το προσωπικό του συνεργάτες μας που ασχολούνται με τους τριμερείς, ε, με τους συνεργάτε <clears throat> διαλόγους, τους συνεργάτες μας από τη γραμματεία. Μερικά από όσα γίνονται τώρα δεν θα πρέπει να τα θέλουμε δεδομένα, διότι πραγματικά ω Επιτροπή έχουμε αναλάβει μερικά τα μείζωνα ζητήματα της εποχής. Ακόμη και για την προστασία των δεδομένων βλέπετε πόσο μεγάλη προσοχή έχει λάβει το θέμα και πόσο ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί σε όλε τι λεπτομέρειε. Ευχαριστώ λοιπόν του συναδέλφου που έχουν ασχοληθεί με τα θέματα αυτά και το προσωπικό του συνεργάτε που τα παρακολουθούν ε, για τι ερωτήσει που τέθηκαν προ τον κύριο Κίρκοπ και αυτό που σχολιάσατε. Βεβαίω, όσο προχωρούν οι τριμερεί διάλογοι, θα σα ε, κάνουμε πιο συγκεκριμένε ερωτήσει. Θα περνάμε και στι λεπτομέρειε των διαφόρων ε, ζητημάτων. Ακόμα λοιπόν, βρισκόμαστε στι πρώτε μέρε του τριμερού διαλόγου. Θα εντατικοποιηθεί ο ρυθμό όσο περνάνε οι μέρε. Ξεκινάμε, ολοκληρώνουμε, μάλλον, ολοκληρώνουμε νωρίς σήμερα. Θα σας δώσω ραντεβού αύριο στις 9. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι.